Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι συζητήσει σχετικά με τις περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 του κανονισμού. Η πρώτη μας συζήτηση έχει ως θέμα την κατάσταση στην Τουρκία και ιδίως την απομάκρυση εκλεγμένων δημάρχων. Πριν κηρύξω την έναρξη αυτής της συζήτησης, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Ολομέλης αυτή τη βδομάδα δοκιμάζεται η λειτουργία ενός νέου συστήματος που επιτρέπει στους βουλευτές να εγγράφονται ηλεκτρονικά για τη διαδικασία Catch the Eye και για τη διαδικασία ερώτησης με τη γαλάζια κάρτα. Έχετε ήδη λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του συστήματος και στα έδρανά σας υπάρχουν και οι σχετικές γραπτές οδηγίες. Μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας για παρέμβαση στη συζήτηση χρησιμοποιώντας τα ειδικά πλήκτρα στο μηχάνημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σημειώστε επίσης ότι παράλληλα με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να υποβάλλετε το αίτημά σας με τη συνήθη πρακτική, δηλαδή υψώνοντας ένα λευκό φύλλο χαρτιού ή υποβάλλοντας αυτοπροσώπως το αίτημα κατά την έναρξη της συζήτησης του συναδέλφου της Ολομέλειας για, τη δικασία, για την διαδικασία Catch the Eye και υψώνοντας μια γαλάζια κάρτα για τη διαδικασία της ερώτησης μέσω της γαλάζιας κάρτας. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια διαφόρων συζητήσεων. Γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να έχετε πάντα μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό θα δοκιμαστεί και στη διάρκεια της συζήτησης που ξεκινά αμέσως τώρα και όπως προείπα είναι η κατάσταση στην Τουρκία και ιδίως η απομάκρυση εκλεγμένων δημάρχων. Δίνω το λόγο για δυόμιση λεπτά στον πρώτο εκ των συντακτών, τον κύριο Λαγκοντίνσκι. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Αγαπητοί συνάδελφοι, αν μπορώ να σας δώσω μια συμβουλή, πηγαίνετε να τράγωνο πιο πέρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να παρακολουθήσετε την ακρόαση. Εγώ την ε, παρακολούθησα χθε. Εκεί μιλάμε για ανθρώπους ε, και για την ελευθερία τους. Εκεί μπόρεσα να δω τη γυναίκα του Ντεμιρτά που αγωνίστηκε για τον σύζυγό τη Σήμερα όμως δεν συμμετάμε τον Ντεμιρτά. Συζητάμε τέσσερις δημάρχους από την Τουρκία, οι οποίοι καθαιρέθηκαν παρότι έχουν εκλεγεί δημοκρατικά ε, έχουμε λοιπόν τους ε, τρεις αυτούς δημάρχους, Μικράτς, Τούρκ ε, και Ερτάν, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εντελώς χωρίς λόγο συλληφθεί τον κύριο Καφτανσιόγλου επίσης, ε, τον ε, πρόεδρο του ΤΕΧΑΠΕ, που επειδή έχει γράψει ένα tweet το 2012, ε, καταδικάστηκε κι αυτός. Και σήμερα μιλάμε και για την ασφάλεια των περασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το ψήφισμα, οι οποίοι οι υπερασπιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, διακινδυνεύουν την ελευθερία και την ε, δική του ε, ακαιρεότητα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα. Επειδή κάποιοι θεωρούν ότι, παραδείγματο χάρη, ένα δικηγόρο εξήβρισε τη δικαιοσύνη, πρόσβαλε τη δικαιοσύνη, ένα δικηγόρο. Και υπάρχουν πολλά άλλα θέματα τα οποία διακυβεύονται πέραν αυτών. Έχει να κάνει το θέμα με τι σχέσει μα με την Τουρκία, το μέλλον των σχέσεών μα. Πώ το βλέπουμε ε, με τη χώρα αυτή. Είναι δύσκολο ε, το μέλλον. Όμως δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το 20% των κρατουμένων στις φυλακές της Τουρκίας να βρίσκονται εκεί λόγω καταγγελιών ε, περί τρομοκρατίας που δεν είναι ε, βάσιμες, που δεν είναι τεκμηριωμένες οι καταγγελίες. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει ακόμη και με την τουρκική κυβέρνηση να έρθουμε σε αντιπαράθεση, διότι δεν μπορούν να στερούν ε, την ε, ελευθερία. Πρέπει να αγωνιστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ανθρώπων και στην Τουρκία. Μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας εδώ, αλλά θεωρώ ότι την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας θα πρέπει να την υπερασπιστούμε και στο μέλλον, όμως ε, πάνω σε μια κοινή βάση η οποία δεν μπορεί να είναι παρά ο αλληλοσεβασμός, αλλά κάτι ακόμη πιο σημαντικό, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόμενο του ψηφίσματος συντάκτης ομιλητής βλέπω στη λίστα ότι είναι ο κύριος Μάντισον αλλά δεν τον βλέπω παρόντα επομένως δίνω το λόγο στον κύριο Σάντσες Αμόρ για 1,5 λεπτό. Thank σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ε, πως εύκολα καταλήξαμε σε συμφωνία με τι άλλε πολιτικέ ομάδε για το ψήφισμα αυτό και αυτό διότι έχουμε πολύ σοβαρή υποβάθμιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ε, Τουρκία και άρα δύσκολο να βρεθούν άλοθη για την Τουρκία. Το ποινικό σύστημα στη χώρα αυτή ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιούν για να μην πω ότι το έχουν σχεδιάσει πολλέ φορέ για να καταστήλουν, για να φημώσουν ε, την πολιτική κριτική ε, οι θύνοντε εκεί. Ε, βλέπουμε τι γίνεται στην κυβέρνηση, τι γίνεται στη διοίκηση, ότι καθερούνται και υποκαθίστανται από μη εκλεγμένου ε, ουσιαστικά υποστηρικτές του κατεστημένου, του ε, κυβερνώντος ε, κόμματος. Μιλάμε για πάυση προσφάτως εκλεγέντος Δημάρχο από την κυβέρνηση από ένα κόμμα ανταγωνιστικό, αντίπαλο και αντικαταστάθηκε ο δήμαρχος από δήμαρχο του ίδιου αυτού κόμματος. Επομένως δεν υπάρχει καμία, κανένα εχέγγυο, καμία εγγύηση και αυτό γίνεται και με το Σοσιαλδημοκρατή Δήμαρχο τη ε, Κωνσταντινούπολη. Δύο φορέ χρειάστηκε να εκλεγεί, να περάσει δηλαδή την εκλογική βάσανο και να επιβεβαιωθεί η εκλογή του. Δεν μιλάμε τώρα για κομματική αλληλεγγύη. Το λέω ξεκάθαρα. Εδώ υποσπερζόμαστε την δημοκρατία ε, στην Τουρκία, ανεξαρτήτω ε, του σε ποια παράταξη πρόσκυνται οι δήμαρχοι. Πολλά πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη χρήση ε, του επιχειρήματος της ασφάλειας, της ασφάλειας, ε, ουσιαστικά για την καταστολή και για τον έλεγχο της τοπικής κοινωνίας. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει η κυρία Αλς Σαχάνη για 1,5 λεπτό. Bästa talman, ärade kollegor. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία την οποία επέδειξαν. Νομίζω ότι οι συζητήσεις που προηγήθησαν ήσαν καρποφόρες και γι' αυτό έχουμε μπροστά μας ένα ψήφισμα το οποίο δεν ασχολείται μόνο ότι ο εκπρόσωπος του Τσέχαπε που κέρδισε κάποιες τοπικές εκλογές ε, Παρ' όλα αυτά καταδικάστηκε σε 8 και σε 9 χρόνια για κάποιες αναρτήσεις ε, του παρελθόντος εντελώς αδικαιολόγητες. Το συγκεκριμένο ψήφισμα υπογραμμίζει τις ανησυχίες τις οποίες έχουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των ε, προβλημάτων που αντιμετωπίζει η δημοκρατία στην Τουρκία υπάρχουν καταχρήσεις της αντιτρομοκρατικής ε, γίνεται μάλλον κατάχρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, κάτι το οποίο είναι ένα στιγμίο το οποίο σημείο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε στις εξωτερικές σχέσεις που έχουμε. Εμείς λοιπόν είμαστε διατεθειμένοι να θέτουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη όταν ε, τίθενται σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και όταν δεν γίνονται σεβαστοί οι κανόνες της δημοκρατίας. Ελπίζω λοιπόν το ψήφισμα αυτό να γίνει δεκτό χωρίς προβλήματα και ελπίζω να υπάρξουν δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, υπήρξαν πράγματα, δημοτικέ εκλογέ στην Τουρκία, ψήφισε ο κόσμο, αποφάσισε και τι έγινε τελικά οι εκλεγμένοι δήμαρχοι δεν μπόρεσαν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. πάυθηκαν, ε, καθερέθηκαν. Αυτό είναι μη δημοκρατικό, είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να το πούμε απερίφραστα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνηση του ΑΚΠ ε, όλο και πιο ε, έντονα στρέφεται κατά της αντιπολίτευσης, κατά του κύριου Καφτανσιόλου από το ΤΣΕΧΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη και για κάποιες αναρτήσεις που έκανε πριν από χρόνια τον καταδικάζει σε σχεδόν 10 χρόνια χρόνια φυλάξη. Αυτό είναι επίση απαράδεκτο στην Τουρκία πάνω από 5.000 μέλη του ΧΑΝΤΕΠΕ είναι πίσω από τα κάγκελα, δημοσιογράφοι, αντιπολίτευση, επικριτές κυβέρνησης ε, είναι φυλακισμένοι ε, και πολύ πολιτικοί όπως βέβαια ο Ντεμιρτάς, στον οποίο θέλω να εκφράσω την πλήρη αλληλεγγύη μου. Ε, επίσης διώκονται αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ερντογάν αυτό που κάνει δεν είναι επίδειξη ισχύω, αλλά επίδειξη αδυναμίας ουσιαστικά με όλα αυτά που κάνει. Η αντιπολίτευση επομένως ε, αντεπιτίθεται και ενδεχομένως κάτι μπορεί να αλλάξει τώρα στην Τουρκία. Αλλά δεν είναι θέμα μόνο του κράτου δικαίου. Έχουμε την ελευθερία έκφραση, την ελευθερία γνώμης που είναι σε κίνδυνο στην Τουρκία. Πολλά διακυβεύονται. Έχουμε τις περισσότερες δολοφονίες γυναικών ε, στην Τουρκία. Αυξάνονται τα νούμερα, βιασμοί, παιδιά ε, σε θρησκευτικά ιδρύματα βιάζονται και ε, πολλές εργαζόμενες σε υποτιθέμενα επαγγελματικά ατυχήματα χάνουν τη ζωή τους. Συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις καταστέλλονται. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το προσέξουμε. Περνάει από μια οικονομική και πολιτική κρίση η χώρα αυτή την περίοδο ο πληθυσμός ε, ζει όλο και χειρότερα. Ε, γι' αυτό λοιπόν ε, τους επόμενους μήνες θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα ακόμη περισσότερο στην Τουρκία και να ξεκινήσουμε με τη δική μας πολιτική αγαπητοί συνάδελφοι, να αφήσουμε την υποκρισία, να αλλάξουμε κι εμείς πολιτική. Έχουμε αυτή το σύμφωνο μετανάστευσης. Βλέπουμε όλο και περισσότεροι όμως να έρχονται από εκεί εδώ γιατί δεν μπορούν εκεί να επιβιώσουν. Το λόγο η κυρία, έχει η κυρία Σόιντροβα για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεργάστηκαν για να κατατεθεί το συγκεκριμένο ψήφισμα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι υποστηρίζουμε έμπρακτα την δημοκρατία και τις δημοκρατικές δυνάμεις στην Τουρκία. Η στάση της κυβέρνησης έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια η κατάσταση των Κούρδων περιπλέκεται όλο και περισσότερο, είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στο παρελθόν. Απαιτείται να υπάρξει δράση από πλευράς μας. Οι εκκλήσεις τις οποίες έχουμε απευθύνει προς την τουρκική κυβέρνηση δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι μεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία αλλά δεν συμπεριφέρεται σαν τέτοιο. Ε, οι οργανώσεις οι κουρδικές μάλλον θεωρούνται στην Τουρκία από την τουρκική νομοθεσία ως τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι διώξεις ε, εις βάρος των Κούρδων πολιτικών είναι συνεχείς και ευρύτατες και συνεπώς κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε μια νέα μορφή γενοκτονίας. Πρέπει να βρεθεί μια λύση και για το κουρδικό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση αυτή Βλέπουμε εδώ ποιοι είναι οι δήμαρχοι οι οποίοι εμποδίζονται στο να ασκήσουν το λειτουργήμά τους. Το θέμα δεν είναι βέβαια μόνο κάτι το οποίο αφορά αυστηρά τους Κούρδους, ε, το θέμα είναι ευρύτερο. Ε, δεν μπορούμε να το ανεχτούμε πλέον, δεν μπορούμε να συνηθίσουμε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Ο Ερντογάν θα πρέπει να κατανοήσει ότι η αντιπολίτευση σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές έχει το δικαίωμα να κερδίζει εκλογές. Λοιπόν, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ασχολείται αυτή τη στιγμή με την Τουρκία και αν δεν αντιδράσει το Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα την... των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει ο κύριος Χριστοφόρου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια κατέστην κανόνα η βία, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η τρομοκρατία εντό και εκτό Τουρκία. Και είμαι εξ που πιστεύω ότι απλώ το θέμα με την παραβίαση των νόμων και των κανόνων για τους εκλεγμένους δημάρχους είναι μια συνέχεια πολλών άλλων παραβιάσεων που μετέτρεψαν την τουρκία σε μια ανοιχτή χώρα φυλακής βίας και τρομοκρατίας μιας τρομοκρατίας η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην τουρκία αλλά εξάγεται και στις γειτονικές χώρες. αγαπητέ κύριε πρόεδρε η χώρα η δικιά μου ολόκληρη υφίσταται τη βία την τρομοκρατία τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων των σκληρών πρόσωπων της Τουρκική επεκτατική κατοχικής τουρκίας εδώ και 45 χρόνια στην κύπρο. είναι γι' αυτό που σήμερα αν πραγματικά θέλουμε να συμβάλλουμε όχι με μόνο ακόμα ένα ψήφισμα αλλά με πραγματικό έργων ως ευρωκοινοβούλιο και ως δημοκρατικά εκλεγμένοι πρέπει να βροντοφωνάξουμε και να στείλουμε το μήνυμα με συγκεκριμένα μέτρα μηδενική ανοχή στην τουρκία εδώ το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και η ευρωπαϊκή ένωση έλαβαν συγκεκριμένα μέτρα για άλλε χώρε και τη ευρωπαϊκή ένωση και εκτό ευρωπαϊκή ένωση χωρί να οροδεί εφαρμόζοντα αρχέ και αξίε. δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε εκτόσει και υποχωρήσει απέναντι στην τουρκία και αν θέλουμε πραγματικά να το καταστήσουμε πράξη οφείλουμε όλοι εμεί οι οποίοι φαντάζομαι κανένας από εσάς δεν ανέχεται να υφίσταται η χώρα σας αυτό που υφίσταται η δικιά μου χώρα αλλά και αυτές οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προχωρήσουμε στον πάγωμα των ενταξιακών κονδυλίων της τουρκίας. κανένα ευρώ σε αυτήν τη χώρα που τρομοκρατεί εντός και εκτός τουρκίας καμία στήριξη καμία βοήθεια καμία ουσιαστική συμπαράσταση προς όλους αυτούς οι οποίοι πραγματικά δημιουργούν πρόβλημα και αστάθεια εντός και εκτός τουρκίας. πιστεύω ακράδαντα ότι και αυτό το ψήφισμα δεν πρόκειται να συγκινήσει τον κύριο Ερτογάν. Ο κύριος Ερτογάν εξαρτιέται σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όσο και αν εκβιάζει και αν απειλεί στην Κύπρο με την παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την καταπάτηση ψηφισμάτων για την αμόχωστο και με τον εκβιασμό για το μεταναστευτικό να ξέρετε έναν κύριε πρόεδρε ότι η τουρκία εξαρτάται σε πολλαπλάσιο βαθμό από την ευρωπαϊκή ένωση και το πάγωμα των κονδυλίων καθώ και το πάγωμα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων είναι αυτό που θα υποχρώσει πραγματικά την τουρκία να ανακρούσει πρίμνα και να σεβαστεί ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών το λόγο έχει η κυρία Σάντος για ένα λεπτό. Έχει, έχουν κλιμακωθεί οι επιθέσεις από πλευρά των τουρκικών αρχών εις βάρος ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών και των γυναικών πολιτικών επίσης. Οι ανησυχίες ε, τον τελευταίο καιρό αυξάνονται και οι διαδικασίες αυτές εις βάρος των τοπικά εκλεγόμενων αρχόντων είναι κάτι το οποίο θα θέσει ακόμα περισσότερο σε κίνδυνο τη δημοκρατία λόγω της απομάκρυνσής τους και της αντικατάστασής τους. Εξελέγησαν με πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά παρόλα αυτά αντικαθίστανται από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εκλεγεί. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και προκαλούν τρομερές ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια επιπλέον κόκκινη γραμμή το να ξεπερνούν με τέτοιο σύστημα αυτή την κόκκινη γραμμή είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ανεχόμεθα. θυμόμαστε τι έγινε, ήταν ξεκάθαρη η νίκη του Τεραπέ στην Κωνσταντινούπολη και όμως εξαναγκάστηκε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Οι νόμοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο και μόνο για να φημώνουν αυτούς που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. Για την ομάδα Renew Europe, για ένα λεπτό, η κυρία Στρουγκάριο. Thank you, Chair. I will continue in Romanian. După 17 ani la putere, fundația regimului lui Erdogan începe să se clatine τα θεμέλια του καθεστώτο του Ερντογάν μετά από χρόνια στην εξουσία αρχίζουν να τρίζουν. Όπω είδαμε και στι πρόσφατε εκλογέ, έχασε 7 στι 10 μεγάλου δήμου τη Τουρκία σε καταδίκη των ε, πολιτικών ε, σε φυλάκιση λόγω υποτιθέμενης εξύβρισης ε, ή ε, η καταστολή και η παρενόχληση ανθρώπων που εκφράζουν τις απόψεις τους ε, ή δημοσιογράφων ε, δείχνουν πόσο απεχθάνεται τη δημοκρατία και την ελευθερία έκφρασης και τα δικαιώματα των πολιτών της χώρας του Ερντογάν. Είδαμε την πάυση αυτών των τριών δημάρχων στον Τιγερμπακύρ, το Βαν και το Μαρντίν. Πρέπει να δούμε τι γίνεται ε, με ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και να δούμε και τι σχέσεις υπάρχουν και με οικονομικά συμφέροντα. New Europe, το λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Κούνκε. Tack, herr ordförande. Den eh, europeiska unionen som institution och vi parlamentariker som folkvalda representanter. Ευχαριστώ πολύ Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης πρέπει να πούμε την αλήθεια για το τι συμβαίνει εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια. Για πολύ καιρό στην Τουρκία. Ουσιαστικά πρόκειται για έγκλημα σε βάρος διεθνών συμφωνιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατοντάδες πολιτικοί, δημοκρατικά εκλεγμένοι δήμαρχοι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί ακτιβιστές, οι οποίοι ε, έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να εκφράσουν τη γνώμη τους, έχουν ε, συλληφθεί και κατηγορούνται για τρομοκρατία, ότι είναι εχθροί της Τουρκίας. Η ομάδα των Πρασίνων ενθαρρύνει τι τουρκικέ αρχές ε, να απελευθερώσουν άμεσα και ανεφόρον όλους ε, τους ε, ανθρώπους που κρατούν στις φυλακές χωρίς ε, λόγο, χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί ουσιαστικά τιμηρωμένες καταγγελίες και κατηγορίες. Θα πρέπει να ξέρουν ότι η προσοχή μας είναι στραμμένη στη χώρα αυτή και ότι θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε. Δεν μας έχει δοθεί άλλη επιλογή, αυτό το διδάσκει η ιστορία. Για την ομάδα ταυτότητας και δημοκρατίας το λόγο έχει ο κύριος Ζήμνιοκ για ένα λεπτό συζητήσουμε. Okay. Meine Damen und Herren, in der Türkei spitzt sich die Lage wieder einmal zu. Κυρίες και κύριοι, η κατάσταση στην Τουρκία εντείνεται συνεχώς. Ο Ερντογάν δρά ως απόλυτος ε, αυτοκράτορας, απειλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με νέα κύματα μεταναστών. Κάνει πόλεμο κατά των Κούρδων στην ίδια του την ε, χώρα και τώρα προχωρά σε καθαίρεση δημοκρατικά εκλεγμένων ε, δημάρχων. Ως επίσημος λόγος ε, δίνεται, δίδεται η υποστήριξη του ΠΚΚ Βεβαίως οι δηλώσεις ε, των κυρίων Νταβούτογλου και Γκιουλ μας δείχνουν πως τα πράγματα δεν έχουν καθόλου έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απορρίψει τις ε, απειλές αυτές, αλλά όχι μόνο αυτό. Επιτέλους θα πρέπει να βγάλει τα απαραίτητα συμπεράσματα. Γι' αυτό θα πρέπει η Κομισιόν επιτέλους να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία άπαξ και διαπαντός. Η Τουρκία δεν ανήκει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Το λόγο έχει ο κύριος Ζαχράντιλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη από το 2004 ήμουν μέλος των διακοινοβουλευτικών επιτροπών ε, με την Τουρκία. Ε, σε αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο δεν είμαι πλέον μέλος, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πια. Δεν έχει ενδιαφέρον. Η Τουρκία έχει αλλάξει πια. Η κατάσταση μετά από το πραξικόπημα, την απόπειρα του πραξικοπήματος, και οι εκαθαρίσεις στο στρατό, στον κρατικό μηχανισμό, στα πανεπιστήμια. Η καταστολή γενικά έχει φτάσει σε επίπεδα τα οποία δεν ε, μπορούν να περιγραφούν. Βλέπουμε ότι το καθεστώς συστηματικά επιτίθεται στους δημοκρατικά εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες, κάτι το οποίο θεωρώ απαράδεκτο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε δίκαιοι με την Τουρκία θα πρέπει να αποφύγουμε αυτό το πολιτικό κρυφτούλι. Να τους εξηγήσουμε ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα γίνουν. Ο κύριος Βίλουμψαν για ένα λεπτό. Tusind tak, formand. Kære kollegaer, situationen i Tyrkiet... Καλημέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι απαράδεκτη. Οι Κούρδοι δήμαρχοι παρότι έχουν εκλεγεί απολύτως δημοκρατικά απομακρύνθηκαν. Ο Ντεμιρτάς παραμένει φυλακή και το μοναδικό του έγκλημα σε εισαγωγικά είναι ότι χρησιμοποιεί την ελευθερία έκφρασης η οποία κανονικά του ανήκει εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες πολιτικοί ακτιβιστές είναι στις φυλακές. Η καταστολή πλέον στην Τουρκία δεν μπορεί να συνεχιστεί, ε, ε, πρέπει να υπάρξουν συνέπειες πλέον. Τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν να μας βρίσκουν ουδέτερους. Ε, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Τα δισεκατομμύρια τα οποία έχουμε στείλει στην Τουρκία θα πρέπει να σταματήσουν έως ότου διασφαλίσουμε τον σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι κάτι που αξίζει στον πληθυσμό της Τουρκίας και είναι κάτι που αντιστοιχεί με τις αξίες μας. Μιλτών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ρίσ Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τις 452.321 ε, ψηφοφόρους ε, του East Midlands που ε, ψήφισαν το κόμμα του Brexit. Σήμερα μιλάμε για το καθεστώς δημοκρατίας στην Ανατολική Τουρκία και σε κουρτικές περιοχές και σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό να βλέπουμε να κινδυνεύει στη γειτονική χώρα η δημοκρατία, στη γειτονιά, στη γειτονιά μας της ε, και Υποτίθεται βέβαια ότι συζητούμε για την προσχώρηση της Τουρκίας στη δημοκρατική Ευρώπη. Είναι υποκρατικό. Υποκριτικό επίσης είναι να ζητούμε δίκαιες δημοκρατικές εκλογές ε, σε χώρες όπως η Τουρκία ενώ προσπαθούμε να υπονομεύσουμε τις επιθυμίες των ψηφοφόρων στις χώρες της Ένωσης. Χθε μόλις ε, Βρετανοί ε, βουλευτές από λιγότερο επιτυχημένα κόμματα ζητούσαν περαιτέρω καθυστέρηση του Brexit για να ε, ξεκαθαριστεί η κατάσταση που θα σήμαινε ουσιαστικά να μην γίνει σεβαστή η ψήφος ε, του Βρετανικού λαού. Ένα πράγμα έχει αυτή η Ομοσπονδία να διδάσκει τελικά, ότι δεν τηρεί τίποτα, γιατί παρανομή ενάντια στους εκλεγμένους για δύο λεπτά, το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριος Σόκολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Τουρκία είναι ένα σημαντικότατο γείτονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέραν των οικονομικών σχέσεων, ένα πολύ σημαντικό κρίσιμο θα έλεγα θέμα είναι το θέμα της μετανάστευσης, όπως επίσης και οι επιπτώσεις ε, της σχέσης που έχει η Τουρκία με χώρες όπως η Βοσνία ερζεγοβινη επηρεάζει τα πράγματα στη Βοσνία Ευζεγοβίνη μέσω συγκεκριμένων πολιτικών σχηματισμών και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Κάποια πολιτικά κόμματα στη χώρα, τη Βοσνία Ευζεγοβίνη εννοώ, δεν σέβονται τη συνταγματική τάξη και τις συμφωνίες του Ντέιτον και στην ουσία παραβιάζουν την συνταγματικότητα και τα δικαιώματα μίας από τις εθνοτικές συνιστώσεις της συγκεκριμένη χώρας. Ειδικά για την Τουρκία τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, βλέπουμε την κατάσταση να χειροτερεύει. Η δημοκρατία φύρεται. Το κράτος δικαίου δεν γίνεται σεβαστό. Η συνταγματική τάξη παραβιάζεται και ιδιαίτερα μετά από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016 η κατάσταση χειρο, χειροτερεύσε ιδιαίτερα στον στρατό και στα πανεπιστήμια. Σήμερα έχει έρθει η σειρά των δημάρχων οι οποίοι πολύ απλά στερούνται του δικαιώματος να ασκήσουν την αποστολή τους. Η κατάσταση αυτή δεν είναι καθόλου καλή οι αρχές ε, πάνω στις οποίες ε, δράζεται η δημοκρατία θεωρητικά και στην Τουρκία, το σύγχρονο λαϊκό κράτος του Ατατούρκ δεν υπάρχει πάρα πολύ απλά. Για να μπορέσει λοιπόν η Τουρκία να συνεχίσει να έχει καλές ε, σχέσεις γειτονίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία πρέπει να επανέλθει σε δημοκρατικά επίπεδα. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε την κατάσταση, αν δεν σεβαστεί η Τουρκία ε, το κράτος δικαίου. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Χελανόμα. Ευχαριστώ. Η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός γείτονας από πολιτικής ε, οικονομικής πλευράς και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους πολίτες. Έχω επισκεφθεί την Τουρκία. Και συνάντησα ανθρώπους αισιόδοξου που πιστεύουν στο μέλλον. Βλέπουν ότι είναι δυνατή μέσω της δημοκρατίας, μέσω των εκλογών η αλλαγή. Απ' την άλλη πλευρά όμως ανησυχούν βλέποντας ε, το πώς ενεργεί η κεντρική κυβέρνηση και το πώς συμπεριφέρεται απέναντι σε εκλεγμένους δημάρχους. Η Τουρκία έχει αιτηθεί την προσχώρησή της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μέλος ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και υποτίθεται ότι έχει δεσμευτεί να τηρεί τις δημοκρατικές αρχές. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχθούμε αυτά που γίνονται σήμερα στην Τουρκία, να πάβονται εκλεγμένοι δήμαρχοι, Πρέπει λοιπόν να εγκρίνουμε αυτό το ψήφισμα για να στείλουμε ένα χειρό μήνυμα προς την Τουρκία και προς τους πολίτες της χώρας ότι εμεί στηρίζουμε και στην Τουρκία τη δημοκρατία. Δύο ερωτήσεις. Γιατί το επίπεδο καταστολής δεν μειώνεται στην Τουρκία γιατί έφτασε στον να αντικαθιστά τους δημάρχους μόνο και μόνο γιατί είναι Κούρδοι. Αυτή η καταστολή, αυτή η φρενή της ουσιαστικά καταστολής ε, είναι κάτι το ακατανόητο. Αλλά βέβαια δύο συνάδελφοι είπαν ότι η ελπίδα ξαναγεννιέται. Η Άγκυρα και η Κωνσταντινούπολη έχουν περάσει στα χέρια νέων και μαλιστών ε, φιλόδοξων ε, και μάλιστα και τρία σημαντικά στελέχη του ΑΚΠ εγκαταλείπουν το κόμμα του Ερντογάν. Ο Ερντογάν ανησυχεί και έχει κάθε δίκιο να ανησυχεί και γι' αυτό χτυπάει με τυφλό τρόπο την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να υπερασπιστεί για μια ακόμη φορά τους δημοκράτες στην χώρα αυτή. Ο κύριος ε, Αλφόνση για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το κατεπήγον ψήφισμα για την Τουρκία οφείλεται στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον δημοκρατίας. Η απομάκρυνση των δηματικών αρχών των τριών μεγάλων πόλεων του Κουρδιστάν μόνο και μόνο λόγω της πολιτικής τους κατεύθυνσης είναι κάτι το οποίο εκπλήσει και πρέπει γι' αυτό ακριβώς να αντιδράσουμε πρέπει να βοηθήσουμε αυτός, αυτούς οι οποίοι δίνουν μάχη για τη δημοκρατία. Ε, το πλαίσιο φυσικά είναι ο αγώνας που δίδει ο κουρδικός λαός για την αναγνώριση των ιστορικών του δικαιωμάτων. Η άρνηση του διαλόγου από πλευράς του τουρκικού κράτους για το θεσμικό καθεστώς της κουρδικής περιοχής είναι κάτι το οποίο είναι μια άρνηση της πολιτικής πραγματικότητας. Πρέπει να αποκατασταθεί η τάξη και η Ευρώπη πρέπει να πιέσει γι' αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε για μια ακόμη φορά τις τελευταίες διώξεις ε, τις οποίες ξεκίνησε ο Ερντογάν εις βάρος των δημάρχων. Ε, κατηγορούνται ότι συνδέονται με τις ένοπλες ομάδες του ΠΚΚ και αντικαθίστανται από κυβερνήτες τους οποίους ε, εγκαθιστά το κεντρικό καθεστώς. Εγώ ήμουν δήμαρχος και ξέρω τι πιστεύουν οι πολίτες για αυτούς που εκλέγουν. Λυπάμαι λοιπόν που για μια ακόμη φορά ο Ερντογάν αγνοεί τη λαϊκή βούληση χωρίς να κινδυνεύει να τιμωρηθεί γι' αυτό. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ύπατη εκπρόσωπος για τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής να πιέσει την Τουρκία η οποία δυστυχώς καταστολή και διώξει στην Τουρκία τροφοδοτούν και τον Ισλαμικό φανατισμό. Βλέποντας την έλλειψη ε, προόδου και την κατάσταση την χένουσα στην Βόρεια Κύπρο, λέει ο μιλητής, είναι θέματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχήσουν στην Ευρώπη. Το λόγο έχει ο κύριος Γεωργίου για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που κουβεντιάζουμε για την Τουρκία έρχεται στο μυαλό μου μια εικόνα. Από τη μια ο κύριος Ερτογάν να κρατά στο ένα χέρι τα τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες και στο άλλο χέρι τους εμπορικούς ισολογισμούς της χώρας του μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες και με βλοσιρόν ύφος να απειλεί τους ευρωπαίους πολίτες και αυτοί να παραμένουν σκυφτοί και γονατισμένοι. Όσο δεν αλλάζει αυτή η εικόνα... Συγγνώμη κύριε Γεωργίου, θα ξαναρχίσουμε την ομιλία σας από την αρχή. Δεν υπάρχει από ό,τι με πληροφορούν μετάφραση στα Ιταλικά. Παρακαλώ να ρυθμιστεί αυτό το πράγμα. Ε, και όταν επανέλθει θα σας δώσω το χρόνο εξ αρχής. Είμαστε εντάξει από ό,τι με ενημερώνουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε παρακαλώ να μηδενιστεί ο χρόνος για τον κύριο Γεωργίου. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που μιλάμε για την Τουρκία έρχεται στο μυαλό μου μια εικόνα. Ο κύριος Ερτογάν με βλοσιρόν ύφος να κρατάει στο ένα χέρι τα τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες και στο άλλον του εμπορικού ισολογισμού τη χώρα του με τι ευρωπαϊκέ χώρε και να τα ανεμίζει απειλητικά απέναντι στου Ευρωπαίου ηγέτε και αυτοί να παραμένουν σκυφτοί και γονατισμένοι. Όσο δεν αλλάζει αυτή η εικόνα, η Τουρκία θα διολυσταίνει στον αυταρχισμό. Θα συνεχίζει να κρατά όμοιρον την Κύπρο, να καταστρατηγεί τη δημοκρατία, να περιορίζει τι ελευθερίε, να παραμερίζει και να διώχνει δημάρχου ακόμα και πρωθυπουργού, να διώκει και Τούρκους και Κούρδους, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι διανοούμενοι. Κυρία Φόντερ Λάιεν και λοιποί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλάξτε αυτήν την εικόνα, αν θέλετε και αν μπορείτε, για να τελειώνουμε επιτέλους με όλα αυτά τα ντροπιαστικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λαγός για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Ακούω για δημοκρατικέ ευαισθησίε και για διάφορα τέτοια πράγματα μέσα στην αίθουσα αυτή και βέβαια έχετε απόλυτο δίκιο να μιλάτε για αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, όμω εγώ θα ήθελα να σα μιλήσω ω ένα άνθρωπο που έχω βιώσει αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, έχω εκλεγεί βουλευτή τέσσερι φορέ, τα τελευταία χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όμω πριν από έξι χρόνια υπήρξε μια παράνομη και άδικη δίωξη ει βάρο μα εμένα, του επικεφαλή του κόμματο που τότε ανήκα και άλλων πέντε βουλευτών μπήκαμε στη φυλακή για 18 μήνες και μείναμε εκεί παράνομα μετά από παρεμβάσει του τότε Πρωθυπουργού της χώρας Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με οπτικοακουστικό υλικό το οποίο υπάρχει και το οποίο είναι προς διάθεσή σας σε όποιον έχει αμφιβολίες για όλο αυτόν, με πιέσεις που ασκήθηκαν πάνω σε εισαγγελεί. Αυτά λοιπόν είναι κατάφορε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκλεγμένων βουλευτών. όσο δε αφορά την τουρκία η στάση τη φυσικά είναι απαράδεκτη η τουρκία πρέπει να τιμωρηθεί η τουρκία ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι μέλο τη ευρωπαϊκή ένωση και το πρόβλημα ξέρετε δεν είναι ο ερντογάν στην τουρκία είναι η ίδια η τουρκία. έτσι έχει μάθει να φέρεται και να καταπατά όλε οι διεθνεί συμβάσει και όλου του νόμου κάνοντα μόνο ό,τι αυτή θέλει. Ο κύριος Κεφαλογιάννης για δύο λεπτά η αντικατάσταση των τριών δημοκρατικά εκλεγμένων δημάρχων δεν παραβιάζει τη βούληση των πολιτών των τριών πόλεων της τουρκίας παραβιάζει την ίδια τη δημοκρατία. η τουρκία ιδίως μετά το πραξικόπημα του 2016 ρέπει σε ένα ιδιότυπο αυταρχισμό που δεν συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης. η τουρκία δεν σέβεται τις αρχές του κράτους δικαίου της δημοκρατίας δεν σέβεται τις σχέσεις καλής γειτονίας δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων της όπως παραδείγματος χάρη η αποκλειστική οικονομική ζώνη της κύπρου και της ελλάδος που παραβιάζονται κατάφορα όλο αυτό το διάστημα και η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να λάβει συγκεκριμένη δράση. η ευρώπη επιθυμεί μια δημοκρατική τουρκία στην ευρώπη δεν επιθυμεί όμως η συμπεριφορά μια χώρας που απειλεί την ευρώπη που δεν σέβεται την ευρώπη. με το σημερινό ψήφισμα καταδικάζουμε μια ακόμα αντιδημοκρατική στάση και ενέργεια της τουρκικής ηγεσίας και του κυρίου ερντογκάν προσωπικά. σας ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. σας ευχαριστώ. το λόγο έχει η κυρία ιντσιρ για ένα λεπτό. Herr talman! var jag åhörare på rättegången. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χτε άκουσα προσεκτικά τις ε, κατηγορίες που ε, απίφθηναν οι εκπρόσωποι τη τουρκικής και της κουρδικής κοινότητας εις βάρος των τουρκικών αρχών. Ε, για να το πω κάπως ευγενικά, το νομικό σύστημα στην Τουρκία δεν λειτουργεί με ικανοποιητικό τρόπο. Συν της άλλης, ήδη από το 2018 είναι η χώρα με τους περισσότερους φυλακισμένους και υποδίωξη δημοσιογράφους. Και τώρα ξέρουμε τι συνέβη στο Μαρντίν, στο Διαμπεκύρ και στο Βαν. Μετά από πολλούς μήνες από τις εκλογές οι εκλεγμένοι πλέον δήμαρχοι απομακρύθηκαν. Τα στοιχεία τα οποία μαθαίνω τώρα είναι ότι και άλλοι δήμαρχοι στην επαρχία του Διαρμπεκύρ έχασαν τη θέση τους. Ε, κατηγορήθηκαν για τρομοκρατία ενώ εργάζονται με ειρηνικό τρόπο για την πρόοδο της περιοχής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάρος, μπορεί να βοηθήσει ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Το λόγο έχει ο Μπουχάιτ για ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να δίνει 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ στην Τουρκία μέχρι το επόμενο έτος αντί να διακόψει επιτέλους τις ε, διαπραγματεύσεις. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της λεγόμενης συμφωνίας για τους ε, πρόσφυγες καθώς ε, αυτή δημιουργήθηκε από την αδυναμία και την αδυνα... ανυπαρξία βούλησης να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Τώρα, αν συνεισέφερε αυτό καθόλου στη μείωση των μεταναστευτικών ροών είναι πάρα πολύ αμφίβολο και έχουμε συνολικά 6 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμών και τώρα απειλεί η Τουρκία να αποσυρθεί από αυτήν την συμφωνία. Βλέπουμε τι γίνεται με τους δημάρχους. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος χαίρεται να καταπιέζει τους άλλους μονίμους. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να συρθεί σε αυτό. Οι πολίτες δεν έχουν μαζοχιστικές ε, τάσεις. Λοιπόν, απευθύνομαι σε σας. Σταματήστε αμέσως τις πληρωμές και τις ενταξιακέ συνομιλίες και σταματήστε να συνομιλείτε με τυράννους. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βουέλς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε την ανησυχητική κατάσταση εγώ θα ήθελα να τονίσω όμως την υποκρισία της Ένωσης ε, στα περί ε, ζητήματα. Δημοτικές εκλογές ε, έγιναν νωρίτερα φέτος σε ολόκληρη την Τουρκία με αποτέλεσμα να έχουμε κόμμα της αντιπολίτευσης πρώτο στην Κωνσταντινούπολη. Όμως σε μια συνάντηση στο ΚΑΠΕ είπε ο Ερντογάν ξανακάνουμε την ψηφοφορία γιατί έτσι θεωρούσε ότι θα έλυνε με συνθήκες δημοκρατίας και νομιμότητας τα προβλήματα και εμείς ε, ε, να θυμηθούμε τι είπε και ο Γκίφερ Χόφστατα μια παράδεκτη ε, απόφαση που κάνει την, ε, το και να διολυσταίνει στη δικτατορία και ότι δεν μπορούμε να συστήσουμε μια τέτοια ηγεσία. Έχουμε λοιπόν ε, έναν συντονιστή της διαπραγμάτευσης για το Brexit που λέει αυτά, ενώ στηρίζει ταυτόχρονα τους Lib Dem που κάνουν το συνέδριο τους και εκεί προσπαθούν να, κατα... να καταρρύψουν μια δημοκρατικά εκλεγμένη και μια απόφαση. Η κυρία Χουίτενταλ. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρητικά πολύ είναι οι λόγοι να είναι κανείς υπομονετικός με την Τουρκία. Είναι μια υποψήφια χώρα, έχει δραματίσει σημαντικό ρόλο στη μεταναστευτική κρίση, που είναι μια πρόκληση για τα κράτη-μέλη. Όμως φτάνει κανείς σε ένα σημείο που εξαντλείται η υπομονή του. Πολύ περιμέναμε και ελπίζαμε να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στη χώρα, να υπάρχει μια σταθεροποίηση των δημοκρατικών θεσμών. Μετά το 16 και την απόπειρα πραξικοπήματος πλέον η κατάσταση είναι ανυπόφορη. Το ΑΚΠ δεν δείχνει σε καμία περίπτωση διάθεση να αλλάξει γραμμή πλεύσης. Και αυτά τα επαναλαμβανόμενα νέα από την Τουρκία αρχίζουμε να τα, μην τους δίνουμε και τόση σημασία. Και αυτό με ανησυχεί. Γιατί βλέπουμε την ε, αποσάθρωση των δημοκρατικών θεσμών, βλέπουμε την φήμωση των ανθρώπων που προσπαθούν να εκφράσουν μια διαφορετική γνώμη. Δεν προσέχουμε τόσο πολύ αυτά τα θέματα. Στις οθόνες υπάρχουν κάποια like, υπάρχουν κάποια ε, σχόλια και αυτά τα προσέχουμε πιο πολύ. Βλέπουμε όμως ότι ε, τραβά το σκηνή στα ωριά του Ερντογάν και δοκιμάζει τα, ε, τις αντοχές μας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Η Τουρκία δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα. Είναι μια χώρα που έχει κάνει αίτηση προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια στο πόσο κανείς μπορεί να αποκλίνει από τις δημοκρατικές αρχές και να εξακολουθήσει να, να θεωρείται ότι προχωρά προς τα ένταξη. Η για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει δυστυχώς σε απαράδεκτες αποφάσεις όπως η απόσυρση των δημάρχων μόλις είχαν εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία, ιδιαίτερα όταν είναι Κούρδοι ή κοντά στους Κούρδους στην νοτιοανατολική Τουρκία, αποδεικνύοντας ότι οι ψηφοφορίες για τον Ερντογάν δεν αξίζουν τίποτα. Η δημοκρατία δεν υπάρχει στην Τουρκία. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο κύριος Ντεμιρτάς, είναι στη φυλακή εδώ και τρία χρόνια για πολιτικούς λόγους. Τι δημοκρατία είναι αυτή. Και δεν μας επιτράπει να τον επισκεφθούμε ήδη από το 2016 και μετά. Γι' αυτό λοιπόν και για πολλούς άλλους λόγους ε, τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία απευθύνονται προς την Τουρκία πρέπει να παριλαμβάνουν συγκεκριμένα μηνύματα πρέπει να περικοπούν οι πόροι προς την χώρα αυτή ως υποψήφια χώρα προς ένταξη. Πρέπει να βοηθήσουμε μόνο την κοινωνία των πολιτών. Ο Ερντογάν θα πρέπει να το καταλάβει. Εμείς θα είμαστε πάντα μπροστά του, πάντα θα είμαστε εναντίον της αυθαιρεσίας. Η τουρκική κοινωνία είναι ζωηρή, ζωντανή και δεν θα της γυρίσουμε την πλάτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως μας λέει η ιστορία, η Τουρκία δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι Ευρώπη. Η Τουρκία είναι μια χώρα 80 εκατομμυρίων μουσουλμάνων. Η δημοκρατία και οι ελευθερίες καθημερινά παραβιάζονται από την ε, δικτατορία του Ερντογάν. Η Ευρώπη έχει δώσει δισεκατομμύρια τα τελευταία χρόνια σε μια χώρα που λειτουργεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και συνεχώς ο Ερντογάν απειλεί με πολέμους θρησκευτικού εναντίον των χωρών μας και εναντίον των πόλεών μας μέσα στις πόλεις μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε το θάρρος να πούμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει αμέσως, μα αμέσως, να διακόψει τις διαπραγματεύσεις και τις συζητήσεις για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη. Για δύο λεπτά ο κύριος Φούρλας. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω ακούσει σήμερα πάρα πολλές διαπιστώσεις, πάρα πολλά συμπεράσματα. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα για μέτρα. Είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Τουρκία. Αυτό είναι ξεκάθαρο έχω σχεδόν την ίδια ηλικία με την εισβολή των τούρκων στην πατρίδα μου και σα το λέω πολύ ειλικρινά ω κύπριο Ευρωβουλευτή έχω κουραστεί έχω χορτάσει από φραστική συμπαράσταση από ψηφίσματα τα οποία η τουρκία πετά στον κάλαθο των αχρήστων. είμαστε έτοιμοι ω ευρωπαϊκή ένωση να λάβουμε μέτρα αποφασιστικά διότι είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Ερτογάν. Α το πράξουμε. νομίζω έφτασε η ώρα να το κάνουμε θύμα της πολιτικής αυτής που συζητούμε σήμερα είναι και η χώρα μου. τα τουρκικά γεωτρύπανα αυτή την ώρα που μιλούμε αγνοώντας το δίκαιο και τους νόμους με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού έχουν περικυκλώσει την πατρίδα μου. την ίδια ώρα προχωρούν σε επικισμό της του, αγνοώντας κάθε ψήφισμα των ηνωμένων εθνών. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι αυτή η πειρατική συμπεριφορά δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από κανέναν ζητώ να ενώσετε τις δυνάμεις σας μαζί μας ώστε να πάρθουν μέτρα για να επιφέρουν κόστος στο καθεστώς Ερτογάν. πρέπει επιτέλους να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα στην άγκυρα πως η κάθε παράνομη ενέργεια θα έχει κόστος και αυτό που χρειαζόμαστε είναι συνεργασία και ειρήνη και όχι τουρκικά ανταηλίκια. σας καλώ να σταθείτε στο πλευρό μας λαμβάνοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της τουρκικής πειρατείας στο εσωτερικό της Τουρκίας και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαυρίδης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η καθαίρεση των τριών Κούρδων δημάρχων θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε όλοι μας. Είναι η σημερινή Τουρκία δημοκρατικό πολίτευμα? ανεξαρτήτως απόψεων η απάντηση δόθηκε χτες ενώπιον του ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων. δόθηκε με νομικά τεκμηριωμένη άποψη από την αρμόδια επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του συμβουλίου της ευρώπης η οποία διαπίστωσε ότι στην τουρκία υπάρχει συστηματική αποτυχία ανεξάρτητης και αμερόληπτης δικαιοσύνης. το ερώτημα λοιπόν για μας είναι το εξής μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη η οποία είναι εργαλείο μιας κυβέρνησης και ταυτοχρόνως να είναι δημοκρατία αυτή η χώρα. άρα λοιπόν το καθεστώς Ερτογάν, το οποίο χρησιμοποιεί τη δικαστική εξουσία ως εργαλείο είναι το ίδιο που παρεμβαίνει στη βουλγαρία στη βοσνία αλλά δυστυχώς και στη χώρα μου στο βόρειο κατεχόμενο μέρος της κύπρου το οποίο μάλιστα πρόσφατα επιχειρεί να ισλαμοποιήσει με βάναυσο τρόπο. το ερώτημα λοιπόν για μας και καταλήγω κύριε πρόεδρε άλλο ένα ψήφισμα ή θα προχωρήσουμε σε μέτρα που να έχουν κόστος. ευχαριστώ. σας ευχαριστώ. το λόγο έχει ο κύριος Ολιβιέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόσφατα ο Τούρκος ε, πρόεδρος Ερντογάν σε την απειλή ότι θα αφήσει να χυθεί στην Ευρώπη μεταναστευτικό κύμα. Πληρώνουμε τα ένοχα σφάλματα. Ε, το ότι δηλαδή εκχωρήσαμε σε άλλους την προστασία των δικών ζωτικών συμφερόντων. Ο κ. Ερντογάν βλέπει τον εαυτό του σαν σουλτάνο μια νέα Οθωμανική αυτοκρατορία και ξέρει ότι είναι σε σχετισμό δυνάμεων η πολιτική και ε, τα ξέρουμε αυτά τα ε, που κάνει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, την εχθρική του συμπεριφορά και στάση. Και πολλές φορές ε, δεν ακούει αυτά που λέμε. Είναι υποχείριό του η διασπορά στην Ευρώπη, όμως εμείς στρέφουμε άλλο το κεφάλι. η κατάσταση που βιώνουμε είναι εύγλωτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει την Ευρώπη αυτοκρατορία της αδυναμίας, ιδίως ό,τι αφορά την προστασία των συνόρων. Ουσιαστικά αφόπλησε τα κράτη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχει κάνει έρμεα μιας μεταναστευτικής απειλής την οποία χρησιμοποιεί τώρα ως όπλο μας και καταστροφή ο Ερντογάν. Δεν είναι σφάλμα απλά, είναι καταστροφή. Στο, το λόγο έχει ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, στο ίδιο έργο θεατές με την Τουρκία να προκαλεί και να προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών και εμείς ως Ευρώπη να αναλωνόμαστε σε θεωρητικές διακηρύξεις και ψηφίσματα χωρίς η Τουρκία να συμμορφώνεται στις εκκλήσεις μας. Ποια είναι τα αποτελέσματα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Να αντικαθιστά με διοικητικές αποφάσεις δημοκρατικά εκλεγμένους δημάρχους με τη συνήθη κατηγορία υπόθαλψης της τρομοκρατίας και να τους αντικαθιστά με κρατικά όργανα. Να συνεχίζεται εδώ και τρία χρόνια την παράνομη κράτηση του ηγέτη του Χατεμπά Σελαχεντίν Ντεμιρτάζ. Να φυλακίζει δημοσιογράφους και να ποινικοποιεί κάθε μια αριστεί πολιτική δραστηριότητα να εισβάλλει στην ΑΟΣ κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απειλεί με επικισμό την πόλη της Αμοχώστου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ματζορίνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι σαφές σε όλους και φάνηκε και από τη συζήτηση ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία ζει ένα αγώνα προς την αυθαιρεσία. Η απομάκρυνση των δημάρχων του Διαμπεκύρ, του Βαν και του Μαρντίν ε, δείχνει ότι φοβάται ε, τις αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας ο Ερντογάν, τα πανεπιστήμια, το στρατό και φυσικά ε, τους πολίτες και τις αποφάσεις τους σε επίπεδο τοπικό. Η μεγάλη αυτή χώρα ζει μια μεγάλη δημοκρατική κρίση, ιδιαίτερα θεωρώντας τον σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο τον οποίο παίζει η χώρα αυτή σε διεθνές επίπεδο, έχουμε μπροστά μας μια κρίση την οποία σαν Ευρώπη δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε εμείς να εξαρτώμεθα και επαφιέμενοι στην τουρκική διακήρυξη ενός τμήματος των εξωτερικών μας συνόρων αντιμετωπίζοντας ε, το θέμα των προσφύγων χωρίς καμία δόση ανθρωπισμού. Ε, μπράβο, αγαπητοί συνάδελφοι. Μετά από δεκαετίες παραβιάσεων των δικαιωμάτων, συλλήψεων δημοσιογράφων, που παρεμβαίνουν στα εσωτερικά ζητήματα χωρών όπως η Βουλγαρία γιατί λένε ότι είναι ε, ένας δικτάτορας τελικά ε, ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι παραβιάζονται εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγχαρητήρια. Καλό αργά παρά ποτέ λέει και ο σοφός βουλγαρικός λαός το ξέρουν και αυτοί που είναι στη φυλακή, το ξέρουμε και εμείς ότι εκατομμύρια παίρνει για να κάνει τα ίδια ο Ερντογάν. Εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρήματα φορολογουμένων Ευρωπαίων. Ε, μάλιστα ένα γερμανικό κοντσέρν κάνει κάποιους ε, διαβουλεύσεις αυτή τη στιγμή και συνομιλίες ε, ενώ τον ατμοσφαιρικό αέρα η Τουρκία τον μολύνει χωρίς να σέβεται κανένα κανόνα. Θα δώσουμε όμως και άλλα χρήματα. Υποκριτικό. Μιλητών, προχωρούμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω δεχθεί τέσσερα αιτήματα, γίνονται και τα τέσσερα αποδεκτά. Το λόγο έχει ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο. pane Σας ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να καταδικάσω και να καταγγείλω τη συμπεριφορά σε βάρος δημοκρατικά εκλεγμένων δημάρχων και να καταδικάσω τις ε, κατάφρασες παραβιάσεις των δικαιωμάτων από μια χώρα που έχει υπογράψει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, και Ελευθεριών ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεν σέβεται όμως αυτές τις ε, θεμελιώδεις αξίες. Γινόμαστε μάρτυρες ε, ψευδών κατηγοριών, ε, παράνομων καταδικών και παραβιάσεις των πλέον θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όχι μόνο ελευθερία δίκαιης δίκης ή ελευθερία έκφρασης. Δικαίωμα αυτοδιοίκησης που είναι υποχρέωση δυνάμει της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μπορεί να ασκήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και κράτη, αλλά και ένωση πίεση. The removal of three recently elected... Τρεις ε, δήμαρχοι του ΧΑΝΤΕΠΕ έχασαν ε, τις θέσεις τους ε, σύντομα, ε, πρόσφατα, ενώ είχαν εκλεγεί με μεγάλη διαφορά και βλέπουμε να παρακάμπτεται η τοπική δημοκρατία στις κωδικές περιοχές και να καταστρέφονται οι υποδομές με δωροδοκία και υπεξαιρέσεις και διαφθορά. Πρέπει όμως να γίνει ε, παλαιόν λειτουργικό το κράτος, να αρχίσει να πληρώνει ε, και τα χρέη και τους ε, μισθούς. Εγώ είμαι φίλη του ΧΑΤΕΠΕ, τον Τιγιαρμπακύρ ε, το έχω επισκεφθεί επανειλημμένος και πραγματικά με ε, σόκαρε η στρατιωτικοποίηση της πόλης και το πώς διαχειρίζει την περιοχή το ΑΚΠ. Μιλάμε για στερματοπλέγματα, για μπλόκα, για τεθωρακισμένα. αν ήταν η δική μου πόλη έτσι, Διερωτώ με ή αν προσπαθούσα να πληρώσω απλά το δημοτικό μου φόρο δεν θα ήμουν εξοργισμένη. Χρειάζεται ο λαός στην Διαρμπακύρα ε, αλληλεγγύη. Γι' αυτό λοιπόν θέλω ε, να ε, συνεργαστούμε με τους αδελφούς δημάρχους, να αδελφοποιηθούμε, γιατί χρειάζεται αλληλεγγύη διασυνοριακά. Ο κύριος Πινέντα για ένα λεπτό. Yes. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απομακρύνθηκαν οι δήμαρχοι των τριών κουρδικών πόλεων και φυλακίζονται πολλές φορές οι δήμαρχοι λόγω της πολιτικής τους δράσης. Και όλα αυτά με τη συνενοχή θα έλεγα εγώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, για την φύλαξη υποτίθεται των εξωτερικών μας συνόρων έχουμε δώσει δισεκατομμύρια και εξακολουθεί να θεωρείται υποψήφια χώρα. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιτάει αλλού, γυρνάει την πλάτη όταν η κυβέρνηση του ΑΚΠ επιτίθεται στα δημοκρατικά δικαιώματα και αγνοεί την πλειοψηφία της χώρας θα πρέπει να παγώσουν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία έως ότου σεβαστεί επιτέλους τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εφόσον ε, θεωρεί ότι είναι σημαντικά τα οικονομικά συμφέροντα, πιο σημαντικά από τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων και των Κούρδων, τότε στην ουσία αφήνουμε ελεύθερο τον Ερντογάν. Ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του Catch Διαπιστώνω μια εντυπωσιακή σύμπτωση απόψεων από όλου του ομιλητέ, κυρία Επίτροπε. Περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω και τις απόψεις τη Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια συζήτηση εύθετη χρονικά που επαναλαμβάνει βέβαια τις ανησυχίες που έχουμε εκφράσει και στο παρελθόν για το κράτος δικαίου στην Τουρκία. Οι τοπικές εκλογές τον ε, Μάρτιο και μετά τον Ιούνιο έδειξαν ποια είναι η λαϊκή βούληση και ο λαός της Τουρκίας είναι υπερήφανος ε, και ασκεί τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Αλλά οι αποφάσεις αυτές ε, της κυβέρνησης δεν διασφαλίζουν την ελευθερία έκφρασης, δεν διασφαλίζουν τον σεβασμό της ε, πραγματικής ε, δημοκρατίας και δεν επιτρέπουν στους πολιτικούς να ε, ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Μετά τις εκλογές του Μαρτίου είδαμε ότι ελήφθησαν αποφάσεις από το τουρκικό κράτος όπου στην ουσία ανέρεσαν τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως ε, είπε και ο Επίτροπος Χάν και η κυρία Μογκερίνη, οι αποφάσεις αυτές υπονόμευσαν τις εκλογικές διαδικασίες και δεν διασφάλισαν τον σεβασμό της λαϊκής ψήφου. και δυστυχώς τα πράγματα χειροτέρευσαν τον προηγούμενο μήνα μέσω της απομάκρυνσης ε, των δημάρχων του Διαβεκίρ του Μαρντίν και, του, α, και της τρίτης κουρδικής πόλης. Η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει να εφαρμόζει τέτοια μέτρα τα οποία είναι περιοριστικά της άσκησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Είναι υποχρέωσή της και ως υποψηφίας χώρας και ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε επανειλημμένα εκφράσει στις τουρκικές αρχές ότι συνειδητοποιούμε κάποια θέματα ασφάλειας τα οποία έχουν αλλά παρόλα αυτά αυτά τα προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας δεν πρέπει ε, να τους ε, δίνει την δυνατότητα να εφαρμόζουν τέτοιου είδους αρνητικά μέτρα και τέτοιες αποφάσεις. Δυστυχώς τα θέματα δεν είναι μόνο σε επίπεδο βέβαια τοπικών αρχών, τα προβλήματα και σε επίπεδο δημοσιογράφων, σε επίπεδο πανεπιστημιακών, σε επίπεδο ε, αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλοί φυλακισμένοι αγωνιστές εδώ και τρία χρόνια. Ο Μυρτάς είναι πάντα φυλακή. Η υπόθεσή του συζητήθηκε και στο Δικαστήριο το Ευρωπαϊκό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατηγορείται για εξύβριση ε, του Προέδρου όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση και ο Καφταντσίουγλου. Θα πρέπει λοιπόν να απαιτήσουμε από την Τουρκία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει ως υποψηφία χώρα, τον σεβασμό των δημοκρατικών δικαιωμάτων. Το θέμα δεν είναι μόνο το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας, είναι το είδος της χώρας το οποίο επιθυμούν οι πολίτες της Τουρκίας. Μια Τουρκία με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, μια Τουρκία χωρίς καταστολή, χωρίς διώξεις και μια κοινωνία που θα προοδεύσει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να εργαζόμεθα για να υποστηρίξουμε μια ευημερούσα και ισχυρή Τουρκία σαν βασικός γείτονας εταίρος και όχι μόνο σαν μια υποψήφια χώρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσουμε τους Τούρκους πολίτες που πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να βασίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ έλαβα 7 προτάσεις ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα. Η επόμενη συζήτηση έχει ως θέμα την Μιαμάρ, Βυρμανία και ιδίως την κατάσταση των Ροχίνγκια. Ε, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Τσαρνέσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, είμαι ένας εκ των συντακτών του σημαντικού αυτού ψηφίσματος που είναι διακομματικό. Πριν από αρκετού μήνε ε, συνάντησα ε, την Πρωθυπουργό ε, και συζητήσαμε το γεγονός πως η φτωχή αλλά τεράστια, πιο μεγάλη και από τη Ρωσία χώρα φιλοξενεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που φεύγουν, εγκαταλείπουν το Μιανμάρ. Δεν είναι πρόβλημα μόνο του Μιανμάρ Βερμανίας επομένως αυτό, είναι πρόβλημα και των γειτονικών χωρών. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα αυτό, το ψήφισμά μας είναι σημαντικό και η φωνή μας, οι συμβουλές μας ε, είναι σημαντικά. πρέπει να ακουστούν. Δεν είναι το πρώτο ψήφισμα για αυτό το θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ είναι αρκετό να μιλούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι η θρησκευτική ελευθερία. Για τρία λεπτά ε, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που το σώμα συζητά την κατάσταση των Ροχίνγκια ε, στη ε, Βερμανία Μιανμάρ και ζητά να σταματήσει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία και να αναλυφθεί δράση από την διεθνή κοινότητα. Δεν ξεκίνησε με την έξοδο τον Αύγουστο του 2017 η κρίση. Πάνω από ένα εκατομμύριο Ροχίνγκια πρόσφυγες φεύγοντας από τη βία ε, έφυγαν σε διαδοχικά κύματα και αυτό ήδη από τις τελευταίες δεκαετίες ε, του προηγούμενου, από το 1990. Μιλάμε για γυναίκες, ε, για παιδιά, πάνω από το 40% κατά από 12. Περνάνε μέρες μέσα σε δάση, γέγγιες γυναίκες, μικρά παιδιά, άρρωστοι, ηλικιωμένοι μέχρι να φτάσουν κάπου σε ένα ασφαλές ε, σημείο. Πολλοί βρίσκονται στον καταβλισμό του Κοξ Μπαζάρ. Είναι το μεγαλύτερο στρατόπεδο. Πάνω από 600.000 άνθρωποι ζουν σε 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα μόλις. Για πολλά παιδιά είναι ε, το μόνο μέρος που έχουν γνωρίσει στη ζωή τους ε, και είναι βάλωτα σε ασθένειες. Δεν έχουν πρόσβαση επίσης στην παιδεία. Είναι σπαραξικάρδι όλα αυτά και πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα παιδιά. Το 2018 θυμάστε όλοι ότι η ανεξάρτητη ερευνητική αποστολή των ΗΠΑ διαπίστωσε ε, ότι έχει υπάρξει, ε, έχουν υπάρξει κλίματα κατά της ανθρωπότητας, ίσως και γενοκτονία. Το 18 το 19 στην έκθεσή της μιλάει για συνεχιζόμενη βία, σεξουαλική, λόγω φύλου, ε, βιασμός από συμμορίες, ε, καταναγκασμός σεξουαλική πράξη και από τις στρατιώτες σε βάρος παιδιών, γυναικών και τρανσέξουαλ. Οι αρχέ στη Μιανμάρ όμως δεν ερευνούν σοβαρά ε, τις ε, ραβιάσει αυτές. Ούτε ε, πηγαίνουν να δικαστούν οι θύτες. Μάλιστα ούτε καν δέχονται ότι έχουν γίνει αυτά. Αυτοί οι ισχυρισμοί όμως καταρρύπτονται γιατί υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις και οι διοικητέ των στρατών αυτών που κάνουν αυτές τι αποτρόπε πράξεις παραμένουν στις θέσεις τους δεν μπορεί να μπει πλέον η δερμητική αποστολή ε, στη χώρα. Δεν υπάρχει ε, με την ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών συνεργασία με τη χώρα. Όμω προσπαθεί ακόμη να βοηθήσει για να ε, βελτιωθεί η κατάσταση των δικαιωμάτων. Είναι καιρό να λάβουμε δράση. Το Συμβούλιο έχει επιμηκύνει τα περιοριστικά μέτρα για ένα έτος σε βάρος του Μιανμάρ, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, Και υπάρχει και απόφαση ποινικού δικαστηρίου για έναρξη πρακτική έρευνα για τα εγκλήματα σε βάρος του πληθυσμού των Ροχήν. Και αυτό είναι κάτι θετικό, αν θέλουμε να υπάρξει λογοδοσία. Δεν έρχεται ευθύνη χωρί δικαιοσύνη, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι δράστε των πολύ σοβαρών αυτών εγκλημάτων πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνη. Το λόγο έχει η κυρία Τζιλ για ένα λεπτό. Since hundreds and thousands of Rohingyas were forced out their homes through mass atrocities. Αναγκάστηκαν λοιπόν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ροχίνγκια να καταλήψουν τις αιστείες τους. Ένα εκατομμύριο περίπου ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων σε περιοχές όπως το Κόξες Μπαζάρ. Έχουν φύγει και σε άλλες χώρες όπως το Μπαγκλαντές το 97% των παιδιών από 15 στα 18 δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε σχολείο. Χρειάζεται λοιπόν βοήθεια. Δυστυχώς ε, δεν έχουμε δώσει βάση, δεν έχουμε δώσει την απαιτούμενη προσοχή. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, πρέπει να τερματιστεί η κρίση αυτή. Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε τον Μπαγκλαντές για να αντιμετωπίσει μόνο του αυτόν τον μεγάλο αριθμό προσφύγων. Πρέπει ε, σε συνεργασία με τους εταίρους μας στο ΑΣΕΑΝ να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των Ροχίνγκια έτσι ώστε να ζήσουν κανονικά οι γυναίκες και τα κορίτσια να νιώθουν ασφαλή και γενικότερα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στα σχολεία. Αγαπητοί συνάδελφοι, η τελευταία αποστολή του ΟΗΕ στη Μιανμάρ προειδοποίησε ότι γύρω σε 600.000 Ροχίνγκια που παραμένουν στην Μιανμάρ ζουν υπό την απειλή γενοκτονίας. Τα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τον στρατό συνεχίζονται ατιμόρυτα. Οι Ροχίνγκια στην Μιανμάρ υφίστανται διακρίσεις, δεν έχουν βασικά δικαιώματα γίνονται αυθαίρετες συλλήψεις, ε, δεν υπάρχει ελευθερία μετακίνησης ε, και ιατρική φροντίδα. Ε, έχουν φύγει εκατοντάδες χιλιάδες προς το Μπαγκλαντές, αλλά και αυτοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς υπάρχει υπερπληθυσμός και ανθυγιεινές συνθήκες στις εγκαταστάσεις. Τα παιδιά δεν πάνε σχολείο και υπάρχει πρόβλημα διακίνησης ε, ανθρώπων και σεξουαλικής ε, εκμετάλλευσης. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στη Μιανμάρ για να δώσουν βοήθεια και να παρακολουθήσουν την κατάσταση. Πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη η Μιανμάρ να δώσει υπηκότητα και πλήρη δικαιώματα στους Ροχίνγκια. Πρέπει να διαρευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες και να λογοδοτήσουν οι δράστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σκεφτεί τα εργαλεία που έχει στην διάθεσή της έτσι ώστε το κράτος και ο στρατός να σταματήσουν. Με στοχευμένες κυρώσεις, με πάγωμα περιουσιακών στοιχείων κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει κυρία Ματίας για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Σε σχέση με το ψήφισμα αυτό, και εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί απέναντι στις παραβιάσεις των οποίων δικαιωμάτων σε βάρος ε, των Ροχίνγκια. Να καταδικάσουμε επίσης τη βία σε βάρος γυναικών κοριτσιών. Πρέπει να καταγγείλουμε τα αποτρόπαια αυτά ε, συμβάντα. Δεν αρκεί όμως η καταγγελία, γι' αυτό στρέφουμε στους αδέλφους. Και σας παρακαλώ, αυτό το οποίο δεν έγινε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ψήφισμα, να υπάρξει ε, δυνατότητα για την ειδική συγγήτρια ε, των Ηνωμένων Εθνών να απευθύνει έκκληση και στη διεθνή κοινότητα και ιδίω να ληφθούν μέτρα σε βάρο στρατιωτικών δυνάμεων που έχουν δύναμη λόγω των εμπορικών συμφωνιών και μπορούν έτσι ανενόχλητα και ατιμόρυτα να παρεμβάσουν ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν πραγματικά προνομιακές σχέσεις ε, εμπορικές με αυτή τη χώρα. Πρέπει λοιπόν ε, οι ενωπες να ενδεχθούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά το μηχανή του κόσμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο δημοκρατικό όργανο που ασχολείται όσο εμείς με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που απευθύνουμε έκκληση για να γίνουν έρευνε σε περιπτώσει παρεμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ιδίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πραγματικά μπροστάριδε. Και γιατί το κάνουμε αυτό, Το κάνουμε γιατί μα ενδιαφέρει η μοίρα των εκατοντάδων χιλιάδων αναξιοπαθούντων, ιδίω στη Βυρμανία. Και δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτουμε ψήφισμα για το θέμα αυτό. Είναι το νη στην ιωστή ψήφισμα. Ε, έχουμε εγκρίνει ψηφίσματα βέβαια, αλλά δύσκολα ε, καταλήγουμε σε συμφωνία με το τι θέλουμε να περιλάβει το ψηφισμά. Σε αυτή την περίπτωση συμφωνούμε και θέλουμε διερεύνηση των εγκλημάτων του στρατού της Μιανμάρ πάνω στους Ροχίνγκια. Θέλουμε πραγματικά να επιληθεί κατάσταση, ε, το, το αδιέξοδο που βιώνουν εκατόντας χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς βοήθεια, χωρίς παιδεία, χωρίς ε, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίσης. Αντίθετα, ε, σε φρικτές συνθήκες ζουν σε ένα νησί ή σε ένα κομμάτι γης που τους παραχωρήθηκε από κάποιες άλλες χώρες. Πρέπει να πάψει να επιδεινώνει την κατάσταση και θέλουμε διάλογο Μπορεί και να μην τον θέλει η κυβέρνηση ε, τη ε, Μιανμάρα διάλογο. Πρέπει όμω να συζητήσουμε μαζί του για την ανθρωπιστική κατάσταση των Ροχίνγκια. Γι' αυτό και απευθύνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τα μέσα και τα εργαλεία να κάνει επιπλέον επιτέλους κάτι. Να γίνει η ατμομηχανή, να γίνει η αιχμή του δόρατος ε, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτή την κατάσταση. Προχωρούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρου των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. το λόγο έχει για δύο λεπτά ο κύριο Λέγκα. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από το 2017 πάνω από 700.000 Ροχίνγκα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ε, τις οικίες τους και να γίνουν πρόσφυγες στον Μπαγκλαντές. Ε, οι ένοπλες δυνάμεις ε, της Μιαμάρ εξακολουθούν να τρομοκρατούν ε, το πληθυσμό, δολοφονίες, καταστροφές χωριών. Συνεχώς η κατάσταση δεν αλλάζει και κανένας δεν διώκεται γι' αυτά. Μάλιστα στην περιοχή της πολιτείας Σερακίν έχουν διακοπεί και οι τηλεπικοινωνίες και υπάρχει και πλήρης άρνηση συνεργασία με τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Το 70% περίπου των Ροχίνγκα σε στρατόπεδα στο Μπαγκλαντές είναι παιδιά, χωρίς ελπίδα και χωρίς μέλλον. Εγώ είχα πάει πριν δύο χρόνια στη Μιανμάρ με τη UNICEF. Είδα ότι τα παιδιά των Ροχίνγκα χάνουν το μέλλον τους διότι δεν μπορούν να πηγαίνουν σχολείο. Οι πολιτικοί της Μιανμάρ δεν προστατεύουν τους ε, πολίτες που είναι καταγωγής Ροχίνγκα και γι' αυτό ε, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τους γυρίσουμε τους, ε, τις πλάτες μας. Ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη με το ολοκαύτωμα, επειδή ακριβώς οι λεγόμενοι καλοί άνθρωποι δεν αντέδρασαν, ήσαν παθητικοί μάρτυρες. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε. και Δημοκρατών, το λόγο έχει ένα λεπτό η κυρία Αρένα. Ευχαριστώ τη Δευτέρα οι ειδικοί της αποστολής των Εθνών σε έκθεση τους επιβεβαιώνουν ότι 600.000 ε, Ροχίνγκια ζουν ε, υπό το, την απειλή γενοκτονίας ε, στη Μιανμάρ και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε από τον Αύγουστο του 2018, 700.000 Ροχίνγκια έχουν πάει στο Μπαγκλαντές. Είναι η μειονότητα πλέον διακόμενη στον κόσμο η Ροχίνγκια και είναι η περισσότερη ανιθαγενής, η μεγαλύτερη ανιθαγενής κοινότητα στον κόσμο. Σίγουρα είναι κάτι σημαντικό να καταγγείλουμε αυτά τα εγκλήματα, αλλά δεν αρκεί όμως αυτό. Ε, και αυτό που πρέπει να γίνει είναι και η Ένωση αλλά και η διεθνής ε, κοινότητα ε, πρέπει να πιέσουν να δώσουν λογαριασμό να λογοδοτήσουν για τα όσα κάνουν οι, υπεύθυνοι και ιδίω οι, υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων, οι στρατιώτε αυτοί και οι διοικητέ. θέλουμε να συνεργαστούμε με τη Μιανμάρ για να διευκαθούν τα εγκλήματα κατά τη και να τιμωρηθούν δράσεις. Ευχαριστώ. Renew Europe. Το λόγο έχει ο κύριος Μπένιον για ένα λεπτό. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ροχίνγκια είναι μια εθνοσκευτική ομάδα στην Μιανμάρη, η οποία δεν έχει επίσημο καθεστώς και άρα δεν έχουν δελτία ταυτότητας. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια σύγκρουση η οποία κλιμακώνεται από τον στρατό που ελέγχουν και την ε, κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν εθνικές ε, εκαθαρίσεις, όπως μας λέει ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ και το 2017 έθεσα το θέμα επίσης στην ε, φιλελεύθερη διεθνή. Βεβαίω η στήριξη του Μπαγκλαντές είναι καλοδεχούμενη, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε και το θέμα του περιορισμού των προσφύγων ε, στο στρατόπεδο τους. Θεωρώ ότι Ροχίνγκια θα πρέπει να είναι πολίτες της ε, Μιανμάρ, είναι η πατρίδα τους εδώ και γενιές, δεν μπορούν να δηλώσουν ότι είναι αλλοδαπή. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρέψουν ως πολίτες της ε, Μιανμάρ, να ξαναφτιάξουν τα χωριά τους, να τους ξαναδοθεί η γη τους. Θέλω η κυβέρνηση της Μιανμάρ να εκπληρώσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις για να προστατεύει όλους τους ανθρώπους στην επικράτειά της. Για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών το λόγο έχει η κυρία Μομπάρη και ένα λεπτό. Um, Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, η τραγωδία των Ροχίνγκια ε, γίνεται άλλο ένα ζήτημα άλλη μια ανθρώπινη τραγωδία την οποία ε, πρέπει να προσθέτει στον κατάλογο του ΟΗΕ. Το Μπαγκλαντές αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα των ε, φρικτών πράξεων της γειτονική του χώρας ε, και η διαδικασία ταυτοποίησης των ανθρώπων αυτών σημαίνει ότι 4.500 άτομα έχουν εγκριθεί για να επιστρέψουν στο, στη Μιανμάρ. Ε, με αυτό το αριθμό θα χρειαστούν αιώνε για να επιστρέψει το 1 εκατομμύριο προσφύγων. Και όσοι ταυτοποιηθούν θα πρέπει να θέλουν να επιστρέψουν χωρίς εγγύηση για την ασφαλειά τους. Ο ΟΗΕ πρέπει να λάβει ουσιαστικά μέτρα για να αποκαταστήσει τα ουσιαστικά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των Ροχίνγκια, οι οποίοι ζουν στην πολιτεία Ραχίνε εδώ και πολλούς αιώνες και Βεβαίως ε, αυτοί οι οποίοι διέπραξαν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας πρέπει να λογοδοτήσουν. Στηρίζω λοιπόν αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Καστάλντο. Δεν τον βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Κατά συνέπεια το λόγο έχει η κυρία Ward για ένα λεπτό. Mrs. you Άσε να κάνω και Ναι, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, δεν ε, είχα καταλάβει ότι έλειπε ο κύριος Καστάλτο. Ωραία. Μετά από δύο χρόνια, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει για το ένα εκατομμύριο ροχίνγκια, πρόσφυγες οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά από την βία που υπέστησαν. Η τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επαναπατρισμού μας δείχνει την ανεπάρκεια των συνθήκων επιστροφής. Η κυβέρνηση της Μιανμάρ πρέπει να δημιουργήσει τις απαραίτητες συνθήκες για να υπάρχει ασφαλής επιστροφή. Σύμφωνα με την Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης υπάρχουν ε, ένα εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι επιζούν μόνο χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διεθνή Κοινότητα να δημιουργήσουν ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο για να αντιμετωπίσουν την κρίση και να ζητήσουμε από τη Μιαμάρ να αντιμετωπίσει τις αιτίε, δηλαδή τη συστηματική βία. Δεν μπορεί να υπάρξει ατιμορρησία του στρατού για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τον Ροχίνγκια. Πρέπει να μπορέσει η κοινότητα αυτή να ζήσει και να ανθίσει. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου Αφζάλ και Βατζίντ Χάν για τη δουλειά που έχουν κάνει στο θέμα. Επόμενος εγγεγραμμένος ομιλητής είναι ο κύριος Κιουτσούκ, τον οποίο επίσης δεν βλέπω παρόντα στην αίθουσα. Επομένως το λόγο έχει ο κύριος Μπιέλαν για ένα λεπτό. Mr. Bielan, you have the floor for one minute. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναμφίβολα η μεγαλύτερη σκεφτική ομάδα ε, που διώκεται είναι χριστιανοί. Σε 128 χώρες διώκονται χριστιανοί. Και ελπίζω το κοινοβούλιο μας να προασπίσει τα δικαιώματα και των χριστιανών κάποια στιγμή σε αυτή τη θητεία. Θέλουμε όμω ε, να υπερασπιζόμαστε του χριστιανού και τι άλλε θρησκευτικέ ομάδε. Πρέπει να τι ε, υπερασπιστούμε. Μία από αυτέ είναι η Ροχίνγκια δίωξη τους που ξεκίνησε εδώ και δεκαετίες. Συνεχίζεται όμως ακόμη και σήμερα και αυτό παρά τον ε, εκδημοκρατισμό της Μιανμάρ. Όλοι ελπίζαμε να σταματήσουν οι διώξεις το 2015, όμως πάνω από 700.000 άνθρωποι έχουν εκδιωχθεί ή αναγκαστεί από μόνο να φύγουν από την ε, Βερμανία, ε, Μιανμάρ και όσοι ε, μένουν εκεί διώκονται. Θα μπορούσε λόγω του φυσικού πλούτου της η χώρα να είναι εύπορη και επίσης γεωστρατηγικά έχει μεγάλη σημασία η δραστηριότητα τεράστιων δυνάμεων όπως η Κίνα, η Ρωσία, είπα είναι πολύ μεγάλη όμως η Βερμανία δεν θα μπορέσει να βρει θέση στη διεθνή κοινότητα αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, κυρία Κινίτση για ένα λεπτό. Ο εισαγγελέα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ξεκίνησε τη διαδικασία έρευνας ε, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εις βάρος ε, των Ροχίνγκια. Είναι μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις όπου χτυπούνται κυρίως ε, τα παιδιά και γενικότερα οι ανήλικοι. Πάνω από 100.000 παιδιά βρίσκονται πρόσφυγες στην Μπαγκλαντές και πέφτουν θύματα καθημερινά εκμετάλλευσης. Δυστυχώς ε, δεν έχουν τα παιδιά αυτά ούτε καν πιστοποιητικό γέννησης. Παραβιάζονται τα δικαιώματα ε, των παιδιών, παραβιάζεται η χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, την οποία παρόλα αυτά έχει προσυπογράψει η Βιμανία, το Μιανμάρ. Συνεπώς λοιπόν δημιουργείται μία γενιά θα έλεγα παιδιών φαντασμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τους πληθυσμούς των Ροκίνγκια να ανακτήσουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Ευχαριστώ. Περνάμε στους λόγους του ενός λεπτού. Κύριε Σχέτμαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι την ε, Δευτέρα δημοσιεύτηκε μια έκθεση του ΟΗΕ με πολύ ανησυχητικές ε, πληροφορίες για τους ε, Ροχίνγκια. Η απειλή της γενοκτονίας είναι πλέον οντονότερη από ποτέ. Και λέει ότι η κυβέρνηση Μιανμάρ δεν έχει κάνει τίποτα για να σταματήσει τη βία. Και άρα οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να αναλάβουν ε, συντονισμένες προσπάθειες για να ασκήσουν πίεση στους υπεύθυνου, Θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Και οι ανθρωπιστικοί ε, οργανισμοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ε, Μιανμάρ για να βοηθήσουν τους ανθρώπους και να παρακολουθούν την κατάσταση. Ο κύριος Πόλτσακ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ένα θέμα που το βλέπουμε συνεχώς ε, και το ε, συζητάμε συνεχώς. Ε, διώξαν τους ανθρώπους από τη χώρα. Παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πάνω από 600.000 άνθρωποι κινδυνεύουν είμαστε στα όρια της γενοκτονίας. Απίστευτη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να βοηθήσουμε τον Μπαγκλαντές, την χώρα που φιλοξενεί πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους ε, στην επικρατεία του σε συνεργασία με τον Αζίαν. Βεβαίως, πρέπει να ζητήσουμε άμεση βοήθεια για τους πρόσφυγες, να ερευνηθούν τα εγκλήματα και να ζητήσουμε συντονισμένη δράση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πρέπει να ερευνήσουμε τα εγκλήματα αυτά και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Τώρα ε, τον λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από όταν το, η Μιανμάρ έδιωξε από την επαρχία Ραχίνε πάνω από 750.000 άτομα. Μιλάμε πλέον πάνω από ένα εκατομμύρια ανθρώπους που φιλοξενούνται στο στρατόπεδο προσφύγων Κόξ Παζάρ Εκεί πέρα βεβαίω υπάρχει ο κίνδυνος ε, ριζοσπαστικοποίηση. Η κατάσταση εντό ε, των στρατοπέδων προσφύγων επιδεινώνεται. Πάνω από 500.000 παιδιά δεν ε, πάνε σχολείο. Η προοπτική γρήγορης επιστροφής φαίνεται ότι απομακρύνεται. Είχαμε και την πρόσφατη προσπάθεια επιστροφής 3.500 ε, προσφύγων, αλλά κανείς τους δεν δέχτηκε να επιστρέψει στη Μιανμάρ λόγω των συνθήκων. Επιπλέον, πέρα από την ανθρωπιστική κρίση, έχουμε και μια γενικότερη πρόκληση ασφαλείας. Οπότε θα πρέπει να ενταθούν συζητήσεις για τις ε, προοπτικές ε, των ανθρώπων αυτών να βρεθούν οι δυνατότητες εκπαίδευσης εκεί που βρίσκονται, η πρόσβαση στην υγεία, ο αντίκτυπος στις κοινότητες που φιλοξενούν και βεβαίως η χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ζητά μια βιώσιμη λύση για τους Ροχίνγκια και τις αρχές της Μιανμάρ έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ασφαλείς εθελοντικές επιστροφές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω της εφαρμογής των ε, συνθήκων ε, που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του διαλόγου του ΙΕ που γίνεται στην Γιανγκούν τον Ιούνιο του 2019 υπό την Προεδρία και του Ειδικού Απεσταλμένου της Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με την παρακολούθηση που αφορά τα πάντα εκτός από τα όπλα και τις διμερείς ε, συναντήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει από την Μιανμάρ να συνεισφέρει στην δημιουργία συνθήκων που θα επιτρέψουν την ασφαλή εθελοντική επιστροφή των προσφύγων ε, στις αιστείες τους. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να ζητάμε την λογοδοσία αυτών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε 14 άτομα και θα συνεχίσει να εξετάζει τακτικά τις ε, κυρώσεις αυτές. Επιπλέον και συμπερασματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να απαλύνει τον πόνο των Ροχίνγκια και θα συνεχίσει να είναι σε επαφή με τις αρχές ε, της Μιανμάρ για να επιστρέψουν. Σας ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπη. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για το πέρας της ζήτησης αυτής από ΣΥΑΡ Πρασίνου, S&D, Renew, UNGL και ΕΛΚ. Εδώ ολοκληρώθηκε η συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Επόμενη συζήτηση, το Ιράν και ιδίως η κατάσταση των ε, υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των ε, φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ηθαγένεια. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους συντάκτες. Ε, η κυρία Φωτίγκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θέλω να αποτίσω φόρο τιμής ε, στις κυρίες, ε, στις γυναίκες και τα κορίτσια του Ιράν για το κουράγιο, το σθένο, την αποφασιστικότητα και την επιμονή τους, όχι μόνο ε, στον αγώνα τους για τα δικαιώματα των γυναικών, αλλά και επειδή ε, υψώνουν τα ανάστηνά τους και μιλούν εξ ονόματος όλης της κοινωνίας και κατά του καθεστώτος. ένα από τα σημαντικότερα ε, αντιπολιτευτικά κινήματα, το Εθνικό Συμβούλιο Αντοχής, ε, έχει στην ε, κορυφή του γυναίκα. Πολλές γυναίκες καταδικάστηκαν πρόσφατα σε μακράς διαρκείας ε, κάθυρξη επειδή διαμαρτύρονται για, την υποχρεωτική, για το υποχρεωτικό φόρμα της μαντήλας. Και Επίσης έχουμε ανθρώπους ε, με διπλή θαγένεια, δηλαδή από χώρα της Ένωσης και το Ιράν, που υποφέρουν με την σειρά τους λόγω διώξεων που τους ασκούνται. Ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή τους. Ευχαριστώ. Δυόμιση λεπτά, κύριε Νόιμαν. Αγαπητοί συνάδελφοι, Βλέπουμε πως υπάρχει αυτή η παράδοση την Διεθνή ημέρα της γυναίκας 8 ε, Μαρτίου να στέλνουμε λουλούδια στις γυναίκες. Μια ειρηνική χειρονομία. 8 Μαρτίου φέτος όμως οι γυναίκες ε, στην ε, Τεχεράνη δέχονταν λουλούδια στο μετρό όπου είναι σε χωριστά βαγόνια έτσι και κάποιες γυναίκες έβγαλαν τη μαντίλα και είπαν ότι ελπίζουμε ότι μία μέρα θα μπορούμε να βαδίζουμε δίπλα-δίπλα με μαντίλα και χωρίς. Και βλέπουμε σε ένα βίντεο πως η ε, οι γυναίκε αυτές πραγματικά κατά τη διάρκεια αυτή τη χειρονομία ε, ένιωθαν την ένταση. Ποια ήταν η απάντηση του Καστότος ε, φυλάκιση. Και όχι μόνο αυτό. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία βραβεύτηκε από εμάς με το βραβείο ε, Ζαχάροφ και καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκιση και ραβδισμούς. Ένα πράγμα λοιπόν είναι σαφές. Το καθεστώς απειλείται από αυτές τις γυναίκες και νιώθει απειλούμενο. Ναι. Πράγματι η κατάσταση στην περιοχή είναι πολύ περιπλοκή, αλλά θεωρώ ότι ακριβώς όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά με το καλό και το κακό, να είμαστε στο πλευρό αυτών που υψώνουν τη φωνή τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που σηκώνουν το κεφάλι για να διαμαρτυρηθούν για το διαχωρισμό των γυναικών στο μετρό και παντού στην κοινωνία. Γιατί όταν κάπου αλλού παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε εμείς δεν επιτρέπεται να σοπαίνουμε εδώ μέσα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνυπογράψετε το ψήφισμα αυτό για τις γυναίκες στο Ιράν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένα μισή λεπτό. Η κυρία Γκούτελαντ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε πολλές αναφορές των, του φρικτού θανάτου ε, μιας ε, γυναίκας η οποία αυτοπυρπολήθηκε αυτό αφού είχε συλληφθεί και καταδικαστεί ε, γιατί ήθελα να παρακολουθήσει ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Τόσο φυσικό, τόσο απλό. Τραγική, τραγική κατάληξη για τη γυναίκα αυτή. Αλληλεγγύη λοιπόν, απόλυτη προς και συλληπιτήρια προς την οικογένειά της. Σήμερα συζητούμε τους πρασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και τους φυλακισμένους διπλής ηθαγένειας στο Ιράν. Στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Οι γυναίκες εκείνες που γονίζονται για τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα στο Ιράν είναι φυλακή πολλές μόνο και μόνο γιατί αγωνίζονται κατά της διάκρισης και πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές, ακτιβιστές ε, για το περιβάλλον είναι στη φυλακή μαζί με αυτούς τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών για μήνες, χρόνια ε, και αυτό δημιουργεί φυσικά πάρα πολλά προβλήματα. Σουτούντε, Μοχαμαμπάντι, είναι λίγες από τις περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν πολλοί διπλής ηθαγένειας που κρατούνται. Πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα. Ευχαριστώ. κυρία Ροντρίγκε για να ε, Πρόεδρε, συζητούμε ένα κατεπήγον ψήφισμα για να ζητήσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων των γυναικών ακτιβιστριών που έχουν καταδικαστεί στο Ιράν και την απελευθέρωση των ε, κρατούμενων στις φυλακές του Ιράν που έχουν πλήθα γένεια, Ιράν, Ευρωπαϊκή Ένωση και ζουν δραματικές συνθήκες. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει πρόσβαση. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με δικηγόρους, με συγγενείς. Οι τρεις τελευταίες γυναίκες ε, που καταδικάστηκαν το έκαναν ε, επειδή στις 8 Μαρτίου ε, σε ένα viral βίντεο έβγαλαν τη μαντήλα τους και μοίραζαν λουλούδια και έλεγαν στις γυναίκες «Ε, μακάρι να μπορούσαν στο Ιράν να περπατάνε δίπλα η μια στην άλλη άλλες φορώντας και άλλες μη φορώντας τη μαντήλα ως αποτέλεσμα προσωπικής απόφασης, ελεύθερης απόφασης. Αυτό ήταν το έγκλημά τους το οποίο θεωρήθηκε ε, απόπειρα σε βάρο της δημόσια ασφάλεια. επίθεση σε βάρο τη δημόσια ασφάλεια. 23 χρόνια κάθεξαν η ελάχιστη ποινή, χωρίς να έχουν εγγυήσει, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα ε, επικοινωνίας με δικηγόρο. Πρόκειται για μια συνεχή εκστρατεία παρενόχλησης ε, των ακτιβιστριών, των δικηγόρων που τις περασπίζονται, των δημοσιογράφων που διαδίδουν όλα αυτά. Και αυτές είπαν ότι θα προχωρήσουν γιατί θεωρούν ότι ήδη πάρα πολύ καιρό έχουν περάσει σε μια φυλακή που δεν είναι άλλη από τη χώρα τους. Θέλουν να προασπιστούν την ελευθερία τους, τα δικαιώματά τους, το μέλλον των κοριτσιών τους. Και αυτό λοιπόν ε, πρέπει να το κάνει και το Κοινοβούλιο. Πρέπει να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα. Η Κομισιόν πρώτα απ' όλα για να πει ότι στον πολιτικό διάλογο με, τον, με το Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια πολιτική προτεραιότητα που δεν είναι άλλη από την παράσπιση των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών του Ιράν. Να στείλει επίσης ένα σαφές μήνυμα στις γυναίκες στο Ιράν. Δεν είναι μόνες τους, είναι μαζί τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είμαστε στο πλευρό όλων αυτών των γυναικών που αντιστέκονται και στις φυλακές και στους δρόμους. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, we are Δεν έχουμε καθυστερήσει ευτυχώς πολύ, αλλά παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας. Τρία λεπτά η επόμενη ομιλήτρια Ζόφκο. Δυστυχώς ε, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι ακτιβιστές της δημοκρατίας αντιμετωπίζουν προβλήματα, καταστέλλεται η δραστηριότητά τους και φυλακίζονται αδικαιολόγητα θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απαιτήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά να απελευθερωθούν όλοι ε, οι, υπήκοοι του Ιράν που έχουν και ευρωπαϊκή ε, υπηκότητα ε, να απελευθερωθούν άμεσα. Οι διαμαρτυρίες που έγιναν ήταν ειρηνικές και αφορούσαν το αν θα πρέπει οι γυναίκες να φορούν την ε, Μαντίλα. Καταδικάστηκαν όμως πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν ε, στις διαδηλώσεις αυτές. Η διαφθορά παρόλα αυτά ε, καλπάζει στη χώρα και δεν αντιμετωπίζεται. Βλέπουμε εντελώς δυσανάλογες μορφές τιμωρίας. Οι γυναίκες απλά συλλαμβάνονται επειδή εκφράζουν την άποψή τους. Σε μια άλλη περίπτωση ε, μια γυναίκα ε, ήθελε να δει ε, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν της δόθηκε η δυνατότητα και γι' αυτό έθεσε τέλος τη ζωή της. Υπάρχουν πάρα πολλοί φυλακισμένοι ε, με ευρωπαϊκή υπηκότητα επίσης, διπλή υπηκότητα και δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί η περίπτωσή τους με δίκαιες δίκες. Το Ιράν ε, καταπιέζει ε, τους πολίτες αυτούς, τους Ευρωπαίους αυτούς πολίτες και έχουμε το ηθικό καθήκον, την εθική υποχρέωση να τους υποστηρίξουμε με αποφασιστικό τρόπο. Εμείς είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τους Ευρωπαίους πολίτες ε, όπου και αν βρίσκονται. Το Ιράν είναι και μία από τις ιδρυτικές χώρες των Ηνωμένων Εθνών και έχει επικυρώσει τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες ε, για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην πραγματικότητα όμως δεν τιμά την υπογραφή της η χώρα αυτή και θα πρέπει να καλέσουμε τις αρχές του Ιράν να σεβαστεί τα διεθνώς συμπεφωνημένα επίπεδα προστασίας. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτές τις γυναίκες που τους πολίτες τους Ευρωπαίους που είναι άδικα φυλακισμένοι. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα μισή λεπτό η κυρία Ernst. Κυρίες και κύριοι, Νομίζω είμαι μία από τις λίγες ε, βουλευτίνες εδώ πέρα που γνωρίζω την ε, Νασίνα προσωπικά. Το 2013 μετά την απελευθέρωσή της την γνώρισα. Μετά από τρία χρόνια ξανακαταδικάστηκε και συνελήφθη ξανά το 2018. Το Μάρτιο του 2019 ε, καταδικάστηκε σε 33 χρόνια για το ότι στήριξε τις γυναίκες που έβγαλαν τη μαντήλα. Δηλαδή απέναντι σε τέτοιες ε, αποφάσεις ε, δεν επιτρέπεται να σιωπούμε. Ανεξαρτήτως του τι άλλο συμβαίνει στο Ιράν. Και η διεθνής αλληλεγγύη χρειάζεται σε όλες αυτές τις γυναίκες. Ε, και ας μην ξέρουμε τα ονόματά τους. Και θα έλεγα το εξής στην Ιρανική κυβέρνηση. Δεν μπορεί μονίμως να αποθούμε την πρόοδο του πολιτισμού Μπορεί να την καθυστερήσουμε. Μπορεί να φυλακίσουμε τους εκπροσώπους της, να τη φημώσουμε. Αλλά η ιδέα της ελευθερίας δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Ούτε με νόμο, ούτε δια της βίας. Και αυτό ισχύει γιατί εμείς... Ε, γιατί αυτό μας κάνει ανθρώπους. Και γι' αυτό μιλάμε για πανανθρώπινα δικαιώματα. Είτε είμαστε στη Δρέσδη που είμαι εγώ, είτε στο Ιράν είτε οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, έτσι ανήκει το, σε αυτές τις γυναίκες ανήκει το μέλλον του Ιράν και αυτό δεν θα αλλάξει. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούν οι δηλώσεις των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ. Ο κύριος Σικόρσκι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ε, σαφώς παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα των γυναικών. Και τιμωρούνται πράγματα τα οποία σε εμά δεν είναι εγκλήματα. Παραδοσιακά οι Σιήτες ε, θεωρούσαν αυτούς πιο φιλελεύθερους από άλλα δόγματα. Αλλά σήμερα το Ιράν είναι μια χώρα η οποία ε, εκτελεί μεγάλο ποσοστό των πολιτών της, ενώ το σύστημα της δικαιοσύνης ε, δεν ανταποκρίνεται σε κανένα σοβαρό κριτήριο. Μεσαιωνικοί μουλάδες ε, αποφασίζουν για τις ε, πίνες ανθρώπων που με τη δική μας λογική δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Νομίζω λοιπόν μπορώ να πω πως αν δεν κάνω λάθος η ομοφιλοφιλία τιμωρείται με θανατική ποινή. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να ενώσω την φωνή μου με όλους όσους μίλησαν για να υπερασπιστώ τις γυναίκες αυτές που αποτελούν στόχο του άδικου αυτού συστήματος δικαιοσύνη. Αλλά το Ιράν είναι πλέον και μια γεωπολιτική πρόκληση. Είχαμε την επίθεση την Σαουδική Αραβία και δεν νομίζω ότι τα βλήματα και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη τα έφτιαξαν ε, κάτι κατσαπλιάδες εκεί στα βουνά της Ιεμένης. Ε, τα έδωσε η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε επίθεση σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Έχω λοιπόν την εντύπωση πως ε, το θεοκρατικό κάθεστος προσπαθεί να προκαλέσει τις είπα για να επιτεθούν. Και ελπίζω ούτε είπα ούτε εμείς να ανταποκριθούμε στην ε, πρόκληση γιατί τα έχουμε ξαναδεί που οδηγούν αυτά. Ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, και Δημοκρατών, ο κύριο Πίτσουλα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορούμε να δεχθούμε να φυλακίζεται μια γυναίκα επειδή προσπάθησε να παρακολουθήσει σε ένα γήπεδο, ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ή να καταδικάζονται σε ποινές ε, μεγάλης διάρκειας φυλάκισης γυναίκες που δεν φορούν ε, τη μαντήλα. Και όχι μόνο να φυλακίζονται, αλλά να καταδικάζονται και σε μαστιγώματα. Υπάρχουν πολίτες που αγωνίζονται για έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και είναι και υπήκοοι και της Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν καν να έχουν ε, μία νόμιμη συμπαράσταση, να έχουν ε, την παράσταση δικηγόρου ή τις απαραίτητε ε, φροντίδες στην τροφονικευτή περίθαλψη ή την πρόσβαση στους συγγενείς του σε δικηγόρο. Παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και οι συμβάσεις Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα τονίζουμε στις δεμερείς σχέσεις με το Ιράν. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ομάδας Renew, κυρία Πόριτ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από την εκλογική μου περιφέρεια είναι Ζανίν Ζαγκάρι Ράτκλιφ. Έχει παράνομα φυλακιστεί για πάρα πολλές μέρες ε, δεν της ε, ε, έκαναν ε, δεκτό το αίτημα για δίκαιη δίκη και τελικά δικάστηκε σε ιονή νόμιμες ε, διαδικασίες από ένα ε, ιονή δικαστήριο. Δεν μπορεί να κάνει διεθνείς κλήσεις και την πετάχρονη κόρη της, την Καπριέλα, μπορεί να τη δει μόνο μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει κρατική ομοιρία για την Αζανίν, που μάλιστα έχει κάνει και απεργία πείνας κατά το παρελθόν και έχει απειλήσει να το επαναλάβει συνεχεί, αν συνεχίζουν να τις θερούν τα βασικά θεμελιώδη ε, δικαιώματα. Το Ρίτσαρντ, ο άντρα της πρόσφατα, είπε πως επειδή η κυβέρνηση έχει στην πρώτη ε, προτεραιότητά της τα θέματα του Brexit, έχει ξεχάσει ε, την Ναζανίν. Και τελικά ξεχνάει μέχρι ε, και βασικά πράγματα πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργό. Δεν έχει επισκεφτεί καθόλου το Ρίτσαρντ ε, από τότε που έχει εκλεγεί. Η Ναζανίν όμω δεν είναι μόνη τη. Υπάρχουν και άλλοι υπήκοοι της Ένωσης ε, που ε, είναι φυλακισμένοι, που τους αρνούνται ελεύθερη δίκη. δίκη. Είναι δικό μας καθήκον να, να ε, υψώσουμε το ανάστημά μα και εδώ και στο εξωτερικό. Να στηρίξετε παρακαλώ το κατεπήγον αυτό. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ των Πρασίνων. Ο κύριο Σούρτασουμ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση των γυναικών στο Ιράν είναι ιδιαίτερω ανησυχητική και δεν μπορούμε παρά να το καταγγείλουμε. Μία από τις τελευταίες τραγικές στιγμές ε, είναι ο θάνατος μιας νέας γυναίκας η οποία κινδύνευε να φυλακιστεί για έξι μήνες επειδή προσπάθησε να μπει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ε, ενδεδειμένη ως άνδρας. Ήδη από τον Ιανουάριο του προηγούμενου χρόνου πάνω από 30 άτομα έχουν, ε, συ, ε, έχουν ε, συλληφθεί, βρίσκονται στη φυλακή επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τον υποχρεωτικό μανδύα. Πρόκειται για φυλακίσεις οι οποίες έγιναν με εντελώς αυθαίρετο τρόπο για λόγους διαζυγίου, για λόγους ε, κατάστασης ε, του γάμου τους για λόγους οικονομικούς. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να ε, βοηθήσουν επίσης και αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία στο Ιράν Δυστυχώς ακούγονται τα τύμπανα του πολέμου, δεν είναι μακριά και γι' αυτό θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να ζητήσουμε τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να επιληθούν τα άλλα προβλήματα. Το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από την προσπάθειά μας να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των γυναικών εξ ονόματος ε, της ε, επόμενης πολιτικής ομάδας η κυρία Σαρτόνεα. Όλοι γνωρίζουν ότι οι γυναίκες στο Ιράν μέχρι το 70 ήταν σαν και εμάς, έφαγαν τα ίδια ρούχα και λειτουργούσαν σαν και εμάς. Από το 79 όμως ήρθε το νέο καθεστώς, ήρθε η Ισλαμική Δημοκρατία και τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάστηκαν. Όπως επίσης και οι εθνικές ομάδες γυναικών, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αναγκάζονται οι γυναίκες που παίζουν να φορούν μανδύες. Υπάρχουν όμως πολλές γυναίκες οι οποίες δεν επιθυμούν αυτό το πράγμα και καθημερινά φωνάζουν, κραυγάζουν υπέρ της ελευθερίας τους έτσι ώστε να μην θεωρείται δεδομένη η υποταγή της γυναίκας στη συγκεκριμένη χώρα. Δυστυχώς στις περισσότερες Ισλαμικές χώρες παραβιάζονται με φρικτό τρόπο τα γυναικεία δικαιώματα. Πρέπει να πολεμήσουμε για τις γυναίκες. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε σιωπηλοί. Σα ευχαριστώ. European Conservative. Εκ μέρου του κόμματο των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριο Βασικόφσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ω πρώην ε, πρέσβη τη Πολωνία στο Ιράν, ομολογώ ότι δεν με χαροποιεί ιδιαίτερο ε, το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε αυτή την ε, ε, ακατάλληλη συμπεριφορά των Ιρανικών αρχών. Θα προτιμούσα να, να μιλούμε για την πολιτιστική συνεισφορά του Ιράν στην ανθρωπότητα. Περιμένουμε από το Ιράν σε αυτού του δύσκολου καιρού να διαδραματίσει ένα πιο επικοδομητικό ρόλο στην περιοχή. Περιμένουμε από το Ιράν να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών και, όσους, και όσων διαμένουν ή επισκέπτονται τη χώρα. Επίσης, περιμένουμε από το Ιράν να σταματήσει την πολιτική των ε, αυθαίρετων σύλληψεων και κρατήσεων και να ε, αποφυλακίσει πάρα αυτά και ανεφόρων όλους τους Ευρωπαίους υπηκόους και ιδιαίτερα τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων των γυναικών. Ελπίζουμε τελικά το Ιράν να εγκαταλείψει κάποιες επιθετικές πολιτικές στην περιοχή. Και αν θέλει πραγματικά φιλικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει το Ιράν κατεπηγόντως να αλλάξει την πολιτική του και να τηρήσει τις διεθνείς ε, προδιαγραφές στην πολιτική. Εκ μέρου τη GUNGL, το λόγο έχει ο κύριος Γουάλλας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στο Ιράν ε, με τρόπο που θα ε, πρόσδεται ντροπή στη Σαουδική Αραβία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε κάποιε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίω δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά το να μην μιλούμε για τι παράνομε αμερικανικέ ε, κυρώσει στο Ιράν, σαν να το αποσιωπούμε τελείω, είναι σαν να αγνοούμε την διεθνή κατάσταση των γυναικών ε, και παιδιών στο Ιράν. Γνωρίζουμε ότι οι οικονομικέ κυρώσει που έχουν επιβληθεί από τη ΣΥΠΑ πλήττουν του φτωχού, όπω τα βασανιστήρια πλήττουν τους αδυνάμους. Κυρίως ε, ο άμαχος πληθυσμός πλήττεται από τις κυρώσεις. Γιατί κάνουμε τους πρωταθλητές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όταν δεν καταδικάζουμε, δεν επικρίνουμε καν ε, αποτρόπες οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιρανικού λαού. Κάτι που δείχνει την πολιτική φύση αυτή τη μέρημνα μα για τα πολιτικά δικαιώματα. Σίγουρα το Ιράν έχει γεωπολιτική σημαντική θέση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη χώρα αυτή για να βγούμε από το αδιέξοδο, γιατί είναι και προ το δικό μα συμφέρον. Και φυσικά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο πολιτικά όπλα. Και αν δεν ε, γίνουν δεκτέ οι τροπολογίε που κατέθεσε η Γκουε, θα καταψηφίσουμε το ψήφισμα για το Ιράν. Η κυρία Ντελούση, μία εγγεγραμμένη. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι είμαι στο πλευρό αυτών των θαραλέων γυναικών ε, που διαμαρτύρονται για τα δικαιώματα στο Ιράν. Ε, έχει αποθρασινθεί το Ιράν στις προκλήσεις ε, αλλά και εμείς δεν ανταποκρινόμαστε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν φύγει από την πυρηνική συμφωνία. Ε, ε, Βρετανοί πολίτες απάγονται, φυλακίζονται, υφίστανται βαρβαρότητα. Αυτό είναι ένα πολιτικό παιχνίδι και η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο παγκόσμιος ε, πρωταγωνιστής της συμφωνίας με κάποια κοινικότητα πρέπει να πω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρεγνύει τα ημάτια της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά τι ωφελούν τα λόγια αν δεν επιβάλλουμε κυρώσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα ονόματα οι πολίτες μας που ζουν στην απομόνωση. Η Τζόλι Κίνγκ, Μαρκ Φέρκιν, η Ναζανίν Ζαγκάρι Ράτκλιφ, η Κάιλ Μοκόβιτς και η Νούσα Σούρι και ο Μοράλ Ταχάς. Έχει έρθει η ώρα τώρα να δράσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά η κυρία Εσταράς Φερραγούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά το Ιράν πρωταγωνιστεί σε μια συζήτηση ε, στον κοινό παρονομαστή που είναι παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δημοσιογράφοι, περασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μειονότητες, ανάπηροι, γυναίκες, ακτιβιστές, άτομα με διπλή ηθαγένεια. Όλοι αυτοί ε, διώκονται, ε, υφίστανται βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις, δίκες για να κάνουν τη δουλειά τους και παρενοχλούνται. Ε, και τι κάνουν, υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτές τις απειλές. Ε, είναι πολλές οι περιπτώσεις, ε, ακούσαμε, για βασανιστήρια και για ανθρώπους που υποφέρουν. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην ε, Σαχάρ ε, Κοντογιάρη, ε, τη κοπέλα με τα γαλάζια. Και τι φταίει, τι έκανε, ήταν γυναίκα και της άρεσε το ποδόσφαιρο, ντύθηκε στα γαλάζια, μεταφιέστηκε σε άντρα για να πάει να δει την αγαπημένη της ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο. Αλλά οι ηγέτες και οι άντρες εκεί δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να πηγαίνουν καν στο γήπεδο. Αυτοπυρπολήθηκε ε, μπροστά από το δικαστήριο όταν άκουσε ότι θα φυλακιστεί. Και ποιο είναι το έγκλημά τη να είναι γυναίκα στη χώρα που οι άνδρες ορίζουν τη ζωή των γυναικών και τους θερούν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα και τα πιο βασικά. Ε, πραγματικά μας συγκλονίζει ο τραγικός ε, θάνατος και η τρομερή περιφρόνηση των Ιρανικών αρχών. Από την αρχή της Επανάστασης πάνω από 20.000 έχουν ε, θανατωθεί. Οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα λένε ότι το Ιράν είναι ε, η μεγαλύτερη φυλακή στον κόσμο για τις γυναίκες δημοσιογράφους. Χρειαζόμαστε διαμαρτυρία, καθόλου σιωπηλή. Και η Επίτροπος Τάισεν που έχει ιδιαίτερη ευαισθησία πραγματικά θα μας βοηθήσει να ε, βγάλουμε μια τέτοια κραυγή η βοήθειας. Ε, δεν θα πρέπει να πάει χαμένο αυτό ο θάνατο. Είναι θαραλές, οι ιρανέ είναι πολλέ και είναι αποφασισμένε για να αγωνιστούν, να κατακτήσουν τα δικαιώματά του. Δεν μπορούμε να τι αφήσουμε στη μοίρα του. Αυτέ είναι η πραγματική Ισλαμική Επανάσταση. Και η Ευρώπη θα πρέπει να είναι παραστάτη στον πλευρό αυτών των γυναικών και υπέρ τη συνείδηση. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Γενά. Οι διακρίσει ε, ει βάρο των γυναικών στο Ιράν είναι καθημερινότητα. Όταν μια γυναίκα, όπω η Σαρ Καβαγιαρή, προτιμάει να αυτοπυρποληθεί από το να κρυθεί από, την, από ένα επαναστατικό δικαστήριο μόνο και μόνο γιατί τόλμησε να πάει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, καταλαβαίνετε σε ποιο βαθμό οι γυναίκε ε, δεν απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Μια κοινωνία η οποία απορρίπτει το μισό του πληθυσμού της δεν μπορεί να μεγαλώσει, δεν μπορεί να αναπτυχθεί δεν μπορεί να εξελιχθεί. Δυστυχώ το Ιράν δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όλα τα κράτη τα οποία παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Τότε ο κατάλογο θα ήταν πολύ μακρύ και θα χρειαζόμουν πάνω από ένα λεπτό για να τι αναφέρω αυτέ τι χώρε. Αλλά το Ιράν είναι εταίρο τη Ένωση. Είμαστε πρωταγωνιστέ τη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. σω ορισμένοι θεωρούν ότι είναι περίεργο να μιλάμε για τα δικαιώματα των γυναικών να μιλάμε για μια πυρηνική συμφωνία. Κι όμω το Ιράν πρέπει να κάνει κάτι και εμείς θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε τη μεγαλύτερη αδικία στον κόσμο που είναι ε, να αρνείσαι τα δικαιώματα στο πάνω από το 50% του πληθυσμού σου. Κύριος Μπάνιον, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν πάντα ήταν ε, στοιχείο επίκρισης. Ε, η ελευθερία έκφρασης περιστέλλεται και δεν είναι μυστικό ότι οι αρχές ε, καταπιέζουν τους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η φυλάκιση, οι άδικες ε, δίκες κυριαρχούν κυρίως μεταξύ των εθνικών μειονοτήτων στο Ιράν. Και όμως οι μειονότητες είναι πάρα πολλές, όπως οι Κούρδοι και διάφοροι άλλοι πληθυσμοί. Ε, ο, ο κύριος Ράκλιφ ή η κυρία Ράκλιφ ε, είναι Βρετανοϊρανή. ιρανη ε, επί μήνες είναι σε προφυλάκηση. Καταδικάστηκε για κατασκοπία μετά από μια πολύ σύντομη και άδικη δίκη. Ο Ρίτσορντ Ράτκλιφ τον συνάντησα πρόσφατα στη Γενέβη. Μου φάνηκε καλός άνθρωπος, ακέραιος άνθρωπος, ο οποίο ε, κάνει μια εκστρατεία πολύ θαραλέα για να ελευθερώσει τη γυναίκα του. Πιο σε γεωπολιτικό επίπεδο, το 2018 η ΕΠΑ έφυγε από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν και επέβαλε κυρώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει ακόμα τη συμφωνία. Αυτό δεν ήταν σαφές μήνυμα για το Ιράν. Πάντως, ε, η Ένωση είναι πιθανός φίλος. Εγώ θα ήθελα το Ιράν να ξανασκεφτεί τις πολιτικές του και την προσέγγιση του στα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως στην ελευθερία λόγου και έκφρασης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε τα θεμέλια για εναρμόνιση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό. Το λόγο έχει ο κύριος Ζεγόμ Ριβιέρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα πρέπει να καταδικάσουμε και να στυλιτεύσουμε όλε τι χώρε που καταπιέζουν τι γυναίκε. Σίγουρα και το Ιράν, όπω αναφέρει το ψήφισμα, είναι από αυτέ, αλλά και η Σαουδική Αραβία. Το Πακιστάν. Δεν θυμάστε ε, τις ε, κατά τη Αζία ε, Αμπίμπη. Επίσης, ε, όλες οι χώρε που έχουν ε, θεωρήσει τον Ισλαμικό νόμο τη Σαρία ω θεμελιώδη του νόμου καταπιέζουν τις ε, γυναίκε. Η χρήση του Ισλαμικού νόμου θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της επίκρισή μα. Επίση έχουμε ορίσει, η κυρία Βαντεράρη έχει ορίσει επίτροπο αρμόδιο για την προστασία της, ε, του τρόπου ζωή μα. Ένας, μια βασική του ενέργεια θα μπορούσε να είναι η καταδίκη τη αερίας, ε, για να μην χρησιμοποιείται από καμία κοινότητα στην Ευρώπη. Και ε, αυτό θα ήταν ένα μικρό βήμα, μια μικρή πρόοδος. Είναι καλύτερο από οποιαδήποτε κείμενο. Χωρί όμω να αναφέρουμε το βασικό πρόβλημα, χωρίς, αν το αποσιωπούμε, ουσιαστικά διευκολύνουμε του καταπιεστές των γυναικών σε πολλοί χώρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Κάνκο. Ανάψτε το μικρόφωνο σας, αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σιλάιτ Η, συγγνώμη, η, στο ποδόσφαιρο. Ε, πήγε στο, ποδοσφαιρικό αγώνα και δεν έκανε κακό σε κανέναν. Ε, και να αντιμετωπίζει ποινή κράτηση, ε, φυλάκιση, επειδή ε, αποπειράθηκε να πάει να παρακολουθήσει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Επίση, ε, η Γκαρία σεφάρα είχε πει στον κόσμο ότι μία 29χρονη αυτοπυρπολήθηκε πριν από δύο εβδομάδες μπροστά στο επαναστατικό δικαστήριο τη Θεχεράνη, της στο Ιράν. Ε, άνθρωποι σαν και αυτήν, ε, ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντιμετωπίζουν παρενοχλήσει, εκδιώξει ε, και κρατήσει ε, φυλάκιση. Δεν είναι έγκλημα η προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από τον Ιανουάριο, 32 άνθρωποι συνελήφθησαν και κρατούνται στι φυλακέ επειδή είναι κατά τη υποχρεωτική μαντήλα. Αυτό είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη αξιοπρέπεια των γυναικών. Τα τελευταία τρία χρόνια. 32 ε, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνελήφθησαν, όπως ο καθηγητής Τζαλάλη και άλλος καθηγητής ε, που βρισκόταν σε επίσκεψη ε, στις Βρυξέλλες. Επίσης, είπατε εκπρόσωπος, είπε στις αρχές του έτους, ότι ο διάλογος είναι ο μόνος τρόπος επικοινωνίας, αλλά δεν αρκεί. Και γι' αυτό η 29χρονη Ιρανή έχασε τη ζωή της, ε, αυτοπυρπολήθηκε μόνο επειδή τη άρεσε το ποδόσφαιρο. Άλλοι είναι στι φυλακέ ε, και είναι άρρωστοι, ενώ πολύ περισσότερε γυναίκε ε, βρίσκονται υπό απειλή στο Ιράν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας να παρακαλέσω και πάλι να τηρείτε το χρόνο αγόρευσή σα. Η κυρία Ροντρίγκε Πάλοπ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, θα σας κάνω όλες να υποφέρετε. Αυτό είπε ο δικαστή που καταδίκασε τρεις Ιρανέ ε, για ειρηνική ε, διαμαρτυρία κατά της υποχρεωτική μαντήλας στο Ιράν. Η καταδίκη σε, φυλά... σε φυλάκιση χωρίς εγγυήσεις, με άδικη δίκη και μάλιστα με βασανιστήρια. 32 γυναίκες συνελήφθησαν στο Ιράν και πάνω από 50 άνθρωποι, επειδή είναι ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, υφίσταται διώξεις. Η υποχρεωτική μαντήλα είναι μια σεξιστική διάκριση που χαρακτηρίζει και στιγματίζει τη ζωή εκατομμυρίων γυναικών και κοριτσιών. Δεν υπάρχει πολιτισμό, δεν υπάρχει θρησκευτική πεποίθηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω πρόσχημα για την παραβίαση τη αξιοπρέπεια και των δικαιωμάτων, ούτε για να μα δίνουν, ούτε για να μα δίνουν. Θα θέλαμε να παροτρύνουμε τις Ιρανικές αρχές να ακυρώσουν τις ποινές και να απελευθερώσουν τις αυθαίρετα φυλακισμένες ακτιβίστριες, να διευκολύνουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να προσπίσουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, της διαδήλωσης ε, και της μη διακριτικής μεταχείρισης. Ε, δεν είναι ότι οι γυναίκε που χρησιμοποιούν τι μαντήλε είναι υποταγμένε και οι υπόλοιπε χειραφετημένε. Αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το σώμα μα ω θρησκευτικό σύμβολο ή λάβαρο τη πατρίδα σε οποιαδήποτε γωνιά του κόσμου. Ευχαριστώ. Mr. Patton. ένα λεπτό, κύριο Κάθε μέρα η ε, Ναζαμίν Ζακάρι Ράτφιλ και άλλες Βρετανές ζουν τραγωδίες στο Ιράν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοβούλιο της είναι συνένοχοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έταξε στο Ιράν ε, ότι ε, θα ε, αρθούν οι κυρώσει των ΗΠΑ. 14 μήνες μετά τίποτα δεν έχει γίνει. Και πήγαν οι πεζοναύτες στο Γιβραλτάρ για να πιάσουν το δεξαμενόπλιο που πήγαινε στη Συρία. Όταν ζήτησε υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Ένωση στα στενά του Ορμούς, τις ανήθηκαν. Είναι σαν να βλέπει τον Πινόκιο να θέλει να γίνει πραγματικό αγόρι, ε, βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο λόγια, καμία συνείδηση και όλο απογοήτευση και ε, εξαπάτηση. Και το κοινοβούλιο τι γίνεται. Εγώ είμαι μέλος ε, της αντιπροσωπείας για το Ιράν. Το Ιου, τον Ιούλιο ήρθα στο κοινοβούλιο και ζήτησα επιγόντω να συνεδριάσει η Ιρανική αντιπροσωπεία. Καμία απάντηση. Ε, ε, προσπάθησα ξανά. Καμία απάντηση. Έχουν περάσει 70 μέρε και ακόμα η ε, αντιπροσωπεία για το Ιράν δεν έχει συσταθεί. 70 μέρε που σαπίζουν στη φυλακή όλε αυτέ οι Βρετανέ. Είναι τραγωδία και τα χέρια μας είναι Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Τζόνς. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρία Τέισεν. Οι ζωές των γυναικών ε, απειλούνται σε πολλές διαφορετικές χώρες και το γνωρίζουμε, αλλά στο Ιράν είχαμε ε, τα παραστατικά δικαστήρια που έχουν αυστηροποιήσει πολύ τις ποινές και για ειρηνικές δράσεις διαμαρτυρίας ανώδυνες από γυναίκες υπερασπίστες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για ποιο λόγο, επειδή είναι γυναίκες, επειδή δεν φορούν τη μαντίλα ή το χιτζάπ, επειδή θέλουν να πάνε στο γήπεδο ή προσπαθούν τουλάχιστον, επειδή ε, δίνουν ε, λουλούδια στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και γυναίκες που πολλές έχουν διπλή ηθαγένεια με κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν στοχοποιηθεί με εκτρές συνέπειες, για παράδειγμα δημοσιογράφοι γυναίκες. Ε, στο BBC ε, Πέρσια ε, ανθρώπινα δικαιώματα, οι υπερασπιστές τους ε, δεν έχουν πρόσβαση σε νομική συνδρομή, σε δικηγόρους. Ε, τους συλλαμβάνουν σε ειρηνικέ διαμαρτυρίε στην Πρωτομαγιά. Είναι μακρύ το ψήφισμα με τα ονόματα και μεταξύ αυτών είναι Αζρίν που την ακούσαμε πολλές φορές. Με δρακόντιες ποινές, χωρίς πρόσβαση σε δικηγόρο, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με εξοντοτικές ποινές. Ε, αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά και θα πρέπει να τα καταγγέλουμε και να κάνουμε κάτι. Να σταματήσει το Ιράν και να ε, γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα των γυναικών οπουδήποτε παραβιάζονται. Ευχαριστώ. Thank you. One minute. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο κύριος Γκρούντλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να χαιρετήσω εδώ το θάρρος όλων των υπερασπιστών των γυναικείων δικαιωμάτων στο Ιράν που καταγγέλουν ειρηνικά την συνεχιζόμενη καταστολή που υφίστανται επειδή ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και αρνούνται την υποχρεωτική μαντήλα. Το 2018 στο Ιράν 100 περίπου γυναίκες συνελήφθησαν για τέτοιες δράσεις και ακόμα κρατούνται τουλάχιστον πέντε από τις γυναίκες αυτές έχουν διπλή ηθαγένεια με κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούνται εχθροί του κράτους και δεν έχουν πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ζητούμε λοιπόν από την Ιρανική δικαιοσύνη να αφαιθούν αμέσως ελεύθερες χωρίς όρους. Και τέλος ζητούμε από τα κράτη-μέλη μας που είναι παρόντα στην Τεχεράνη να κάνουν ό,τι μπορούν για να λάβουν τον πλήρη κατάλογο των κρατουμένων που έχουν διπλή ηθαγένεια με κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να τα υποστηρίξουν και να τα προστατεύσουν με επισκέψεις στις φυλακές, με δημόσιες δηλώσεις και ε, διπλωματικά διαβήματα για να ε, αφαιθούν γρήγορα ελεύθεροι. Ευχαριστώ. Κυρία Δεβαλιέρη, ένα λεπτό. Πρόεδρε. Στο Ιράν οι διακρίσεις, οι εκφοβισμοί και οι καταπιέσεις αντίον των γυναικών έχουν αυξηθεί από τότε που οι γυναίκες στο Ιράν αποφάσισαν να, μέσω της, του διαδικτύου να καταγγείλουν τις ε, υπερβολές της ε, αστυνομίας ηθών και τι, τι βασανιστήρια και τι περνάνε κάθε μέρα. Η Ευρώπη βασίζεται στην ελευθερία και στην ευθύνη. Δεν μπορεί να δεχθεί αυτές τι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνονται συστηματικά από ένα πολιτικό σύστημα αρχαϊκό που χρησιμοποιεί την ε, μουσουλμανική θρησκεία για να επιβάλλει την άποψή του. Αυτός ο φανατισμός ε, διαδίδεται και στην ε, Ευρώπη και είναι θύματα οι γυναίκες με αυτή την υποκουλτούρα. με την συνενοχή της αριστεράς. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε και να μην διαδώσουμε και διαφυλάξουμε τις πολιτιστικές μας αξίες. Η αλληλεγγύη της Ευρώπης προς τις γυναίκες του Ιράν θα πρέπει να αφορά όλες τις γυναίκες που είναι μουσουλμάνες και που ζουν και στην Δύση. Γιατί δική μας ελευθερία είναι δική τους ελευθερία και ασφάλεια για όλους μας αύριο. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Ο κύριος Τσαρνέτσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο Ιρανικός λαός έχει μακρά και καταπληκτική ιστορία, αρχαία ιστορία και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πιο απαιτητικοί από το Ιράν σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα των γυναικών. Δεν είναι παράδοξο για έναν λαό με τόσο μακροχρόνια ιστορία. Πριν ε, ε, 40-50 χρόνια ε, με, το Σάχ, με το Σάχ είχαν πολύ περισσότερα δικαιώματα γυναίκε τότε από ότι σήμερα. Υπάρχει παλινδρόμηση, παναχώρηση στα δικαιώματα των γυναικών και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό. Στα θέματα των δικαιωμάτων ε, των ανθρώπων και των γυναικών θα πρέπει ε, να σκεφτούμε και τη φωνή εκείνων που βρέθηκαν στο Ιράν, μετά έφυγαν και μπόρεσαν να, να μας μεταφέρουν αυτά που πραγματικά συμβαίνουν εκεί. Και μάλιστα σε μια διάσκεψη άκουσα τη φωνή γυναικών, μεταξύ άλλων και της κυρίας Ρατζαβή. Θα πρέπει λοιπόν να μην ξεχνούμε όσους μιλούν για το Ιράν και κυρίως όσους έχουν διπλή ηθαγένεια, έχουν και ηθαγένεια ευρωπαϊκή. Θα πρέπει όλους αυτούς τους ανθρώπους να ε, τους έχουμε κατά νου και να μεριμνούμε για το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Κυρία Ρέγνερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών στο Ιράν, το 70% σύμφωνα με μια μελέτη, είναι κατά της υποχρεωτικής μαντήλας. Αυτό το λέει ένα ερευνητικό Ινστιτούτο του ίδιου του Ιράν. Όλο και περισσότερο ε, διαμαρτύρονται οι γυναίκες κατά της ε, καταναγκαστικής μαντήλας για να μπορεί κάθε γυναίκα να αποφασίζει τι θα φοράει, χωρίς να φοβάται ε, την ε, παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Από τον Γενάρη του 2018 ε, δεκάδες γυναίκες και άνδρες έχουν συλληφθεί. Η ειρηνική διαδήλωση είναι ανθρώπινο δικαιώμα και ανήκει σε κάθε κοινωνία. Πολλές ε, θαραλές γυναίκες διαδήλωσαν ειρηνικά κατά αυτής της νομοθεσίας της διακριτικής για την υποχρεωτική μαντήλα και καταδικάστηκαν σε σκανδαλώδεις ποινές 16 έτη κάθεξης μέχρι και 24 έτη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, απαράδεκτα. Ε, απαιτούμε να φεθούν αμέσως ελεύθερες. Thank you. Ευχαριστώ. Κάλμπρο. Κάλμπρο, ένα λεπτό. Πρόεδρε, τους τελευταίους μήνες η κατάσταση στο Ιράν έχει επιδεινωθεί. Όλο και μεγαλύτερη καταπίεση υφίστανται οι γυναίκες. Διάφοροι ακτιβιστές έχουν συλληφθεί γιατί μοίρασαν λουλούδια χωρίς να φοράνε τη μαντήλα. Και μάλιστα πού το έκαναν αυτό, στο μετρό. Ήταν μια απόλυτα ειρηνική κίνηση αυτή. Καταδικάστηκαν οι γυναίκες αυτές σε πάρα πολλά χρόνια φυλάκισης έως και 24 χρόνια. Πρέπει να σταματήσει ε, αυτό το καθεστώς, πρέπει να πέσει αυτό το καθεστώς στο Ιράν. Εμείς θα πρέπει να είμαστε μία φωνή, δυνατή, υπέρ των γυναικών. Όλοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν ελεύθερα το σώμα τους και τη ζωή τους. Βέιμερς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ιδέα ότι μια γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε είναι τραγική. Φανταστείτε να ήταν η αδερφή σας. Φανταστείτε να ήταν κάποιος δικό σας. Μόνο και μόνο γιατί την καταδίκασαν ε, την καταδίκασε κάποιο δικαστήριο. Ο Υπουργό Εξωτερικών ε, του Ιράν δεν συμφωνεί με κάποιες συμπεριφορές στη Σουηδία. Δεν συμφωνεί με το να βγάζουν τις, ε, τη μαντήλα οι γυναίκες ε, στη Σουηδία αν και δεν έχει και τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο αν το κάνανε στο Ιράν. Θα πρέπει με βάση τις δικές μας αξίες να αντιταχθούμε σε ένα βαρβαρικό καθεστώς. Και θα πρέπει να μην δεχόμαστε αυτές τις, αυτά τα, συμβολικά, τα σύμβολα καταπίεσης εναντίον των γυναικών. Κύριε ένα λεπτό. Συνάδελφοι, οι γυναίκες στο Ιράν σε όλους τους τομείς κοινωνίας σχεδόν υφίστανται τεράστιες διακρίσεις. Μεταξύ άλλων αυτό ισχύει και για το νομικό σύστημα στο Ιράν, το σαρί, τη Σαρία δηλαδή, το μουσουλμανικό νόμο που επιβάλλει και τη θανητική ποινή. Το κληρικό δικτατορικό καθεστώς βασίζεται σε ε, πατριαρχία και αποκλεί ε, την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των μειονοτήτων κτλ. Είναι πολλές οι ακτιβίστριες και αυτό ε, δείχνει πόσο ε, κατάπτυστο είναι αυτό το σύστημα. Ε, καταδικάζονται σε ραβδισμού, σε ραπίσματα, σε πολιετή φυλάκιση. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Όσο κυριαρχεί αυτή η θρησκευτική δικτατορία, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ε, για ε, την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Κύριο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω Εκφράζοντα το βαθύτατο σεβασμό μου και την αλληλεγγύη μου προ ε, όλου του υπερασπιστέ ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Με συγκινεί ιδιαίτερω η γενναιότητα των Ιρανών γυναικών που επέλεξαν ένα τόσο φιλερινικό τρόπο για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Μοιράζοντα λουλούδια σε άλλε γυναίκε στον υπόγειο, ε, στο μετρό δηλαδή και συζητώντα τα δικαιώματά του. Σε κάποιο βαθμό μου θύμισε η δική του αντίσταση, τη δική μα φιλερινική αντίσταση στη Σοβιετική κατοχή, ιδιαίτερα με το βαλτικό τρόπο. Εμείς όμως καταφέραμε να διεκδικήσουμε και να ε, κερδίσουμε την ελευθερία μας, ενώ οι Ιρανοί συνάδελφοί μας καταδικάζονται σε απίστευτης διάρκειας ποινές φυλάκισης. Συνεχίζονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι καταπιέσεις, ο εκφοβισμός ε, ε, πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια του Ιράν, κάτι που απειλεί την παγκόσμια ασφάλεια και οικονομία και δημιουργεί μια αστάθεια περιφερειακή. Ζητώ λοιπόν από την Ιρανική, ε, κυβέρνηση να τηρήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και, θεμελιώ, και τις θεμελιώδεις ελευθερίες με βάση τους, διεθνεί τις διεθνείς και τι διεθνείς συμφωνίε που έχει υπογράψει. Και επίση ζητώ από το Συμβούλιο να επαναθεωρήσει τη θέση του για το Ιράν, εξετάζοντα και συμπληρωματικέ κυρώσει. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει η κυρία Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση των γυναικών στο Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολη, δεινή. Θα πρέπει να δίνουν μάχη για τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Ο λιθοβολισμός είναι μια ποινή που προβλέπεται από το Ισλαμικό ποινικό δίκαιο. Ακόμη και όταν είναι θύματα βιασμού ε, τιμωρούνται όπως ε, και ο αυτούργος. Επίσης είναι υποχρεωμένες να φέρουν τη μαντήλα. Νομίζω ότι χρειάζονται κάποια βοήθεια και υποστήριξη στον αγώνα τους. Οι υπερασπιστέ ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γυναικών, ακόμη και με διπλή ηθαγένεια, χωρί να έχουν πρόσβαση σε δίκαιη δίκη καταδικάζονται σε μακροχρόνιες ποινές και πρόσχημα πολλές φορές ε, για την επιβολή ποινών είναι πιθανές επαφές με μη κυβερνητικέ οργανώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή επαφή με τα ΜΜΕ. Και μάλιστα η Ιρανική κυβέρνηση υποτίθεται θέλει να συσφίξει τι σχέσει τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να, την καλέσουμε, να καλέσουμε την Ιρανική κυβέρνηση να τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μην ποινικοποιεί του ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να σέβεται τα δικαιώματα των υπηκών των ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Κουταγιάρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και η γυναίκα είναι ένα ανθρώπινο πλάσμα και έχει αναφέρετα, αναπαλωτρίωτα δικαιώματα. Δεν μπορεί να τα στερείτε αυτά. Εμείς πιστεύουμε στο κράτος δικαίου και γι' αυτό θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες να τη χάνουν παντού προστασία και εντό και εκτός των σύνορων μας. Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της ανεξιθρησκείας, τη θρησκευτική ελευθερία και των πολιτιστικών δικαιωμάτων, αλλά δεν θα πρέπει αυτές οι αρχές να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την ε, δίωξη και την καταπίεση των Ιρανών γυναικών. Κάποιοι ακτιβιστές, ε, υπερασπιστές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπέρμαχοι της ελεύθερης κοινωνίας, είναι δυνατόν να υπόκειται διώξεις για τις πεπιθήσεις τους αυτές. Θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διεθνείς διατάξεις. Θα πρέπει να σταματήσει η άσκηση βίας εις των γυναικών. Θέλω λοιπόν ε, να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με αυτή των συναδέλφων μου και να απευθύνουμε έκκληση προς το Ιράν να σεβαστεί τα δικαιώματα των γυναικών και να αποφύγει τις διακρίσεις βάρος τους. Ευχαριστώ. Η κυρία Ραφαέλ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Τρεις Ιρανές γυναίκες, ακτιβιστές, εξαφανίστηκαν και καταδικάστηκαν σε 16 και 23 χρόνια φυλάκιση. Μόνο και μόνο γιατί αποφάσισαν τι θα φορέσουν. Στην πραγματικότητα είναι ένα καθεστώς ανδρών που τιμωρεί τις γυναίκες ε, που διεκδικούν τα δικαιώματά τους και την ισότητα. Δεν πρόκειται για απομονωμένο γεγονός. Το καθεστώς Να ξεκινήσετε παρακαλώ από την αρχή. Υπάρχει πρόβλημα με κάποια διερμηνία. Θα ξεκινήσω. Από την αρχή. Επίτροπε, Πρόεδρε, συνάδελφοι, τρεις ε, ακτιβίστριες γυναίκες εξαφανίστηκαν και ε, καταδικάστηκαν 16 και 23 χρόνια φυλάκισης. Μόνο και μόνο γιατί αποφάσισαν τι θα φορέσουν μόνες τους. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα καθεστώς ανδρών που φοβούνται τις γυναίκες όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους και ζητούν ε, ισότητα. Και αυτό το τραγικό γεγονό δεν είναι απομονωμένο. Το Ιρανικό καθεστώ έχει μακρά ιστορία παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χιλιάδε ε, ψευτοδίκε έχουν γίνει και ορισμένε οδήγησαν και στη θανατική ποινή. Επίτροπε, σα ε, καλώ εσά και την είπατε εκπρόσωπο να κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτω ώστε να αποκατασταθούν τα δικαιώματα αυτών των θαραλέων γυναικών. Καμία κυβέρνηση θα πρέπει να φυλακίζει και να φυλακίζει γυναίκε μόνο και μόνο γιατί φορούν κάτι που δεν αρέσει το καθεστώ. Ούτε στο Ιράν ούτε πουθενά αλλού. Δεν χρειαζόμαστε του άντρε στην εξουσία να μα υποδεικνύουν τι ακριβώ θα φοράμε. Με ευχαριστώ. Διαδικασία κάτσε τώρα. Mr. Lopez Aguilar. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ για ένα λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, αυτή είναι μια συζήτηση ε, που ήθιστε να κάνουμε την Πέμπτη το πρωί στην Ολομέλεια για τις κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκφράζουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες και τις αρχές της κοινωνίας που εμείς εκπροσωπούμε και αυτό καθορίζει την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Με ένα ψήφισμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση και είναι σπάνιο, ε, είναι ομόφωνο ομόφωνο στην έκφραση της καταδίκης που αξίζει συστηματική και κατάφορη παραβίαση των γυναικείων δικαιωμάτων και η διακρίση εις βάρος τους στο Ιράν. Ε, ακούστηκαν με πολύ ωραίο τρόπο ε, αυτές οι φρικτές περιπτώσεις. Μια γυναίκα αυτοπυρπολήθηκε δραματικά επειδή πήγε στο γήπεδο ντυμένη άνδρας και ήξερε ότι θα καταδικαστεί. Είναι απάνθρωπες ε, οι ποινές αυτές και εξευτελιστικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε μια προσπάθεια για να διατηρήσει τη συμφωνία με τα, για τα πυρηνικά με το ε, Ιράν, με τη διπλωματία, με τις αξίες και τις προτεραιότητες. Αυτό δεν μειώνει, σα ίσα ενισχύει το ηθικό ανάστημα που έχουμε για να απαιτήσουμε κάποια πράγματα για τη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και τη δίωξή τους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, η κυρία Ντέιλι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ πραγματικά είμαι στο πλευρό των γυναικών που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα στο Ιράν. Υποστηρίζω απολύτω την έκκληση να φεθούν ελεύθερε οι γυναίκε που έχουν φυλακιστεί για πολιτική δράση και για τη διαμαρτυρία του για να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα να φοράνε ό,τι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Και καταγγελώ απολύτω και καταδικάζω τη θανατική ποινή και για ανηλίκου. Πρέπει να πω όμω ότι το ψήφισμα δεν είναι ισόρροπο. Αυτή τη στιγμή που είναι σημαντικό το ύφος μας, τη στιγμή που το Ιράν βάλεται και πολιορκείται από πολλού διεθνεί πρωταγωνιστέ. πρωταγωνιστές. Τα ακούσαμε αυτό. Λένε ότι το Ιράν ε, προσπαθεί να προκαλέσει πόλεμο με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Μα οι Ηνωμένε Πολιτείε έσχισαν την πυρηνική συμφωνία και αποχώρησαν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε στραγγαλίζουν την πολιτική του Ιράν και προκαλούν τεράστιο πόνο σε γυναίκε και παιδιά. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξει το Ιράν. Δεν είναι η μόνη και βέβαια πρέπει να αλλάξουν. Και χαίρομαι που τώρα έχουμε ε, στην ε, Ιρανική Βουλή τόσες γυναίκες όσους κληρικούς από την άλλη. Αλλά ε, δεν θα ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα αν δεν συμπεριληφθούν οι τροπολογίες για τις κυρώσεις. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Σκέλη. Συμφωνώ με αυτά που είπαν πολλοί προλαλήσαντες. Η κατάσταση των γυναικών στο Ιράν είναι απαράδεκτη και ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ ήμουνα μέλο στην αντιπροσωπεία με το Ιράν στην τελευταία κοινοβουλευτική θητεία και κάναμε ό,τι μπορούσαμε, ούτω ώστε να διατηρηθεί η πυρηνική συμφωνία. Αλλά θα πρέπει να γίνουν προσπάθειε και ο πλευρά Ιράν, όπω υπόθηκε. Να επιτρέψουν στο Ιράν να ζουν ελεύθερα, γιατί το αξίζουν. Και όπω είπε και ένα βουλευτή ε, οι άντρε στο Ιράν θα πρέπει να λένε στι γυναίκε τι να φορέσουν. Συμφωνώ με την Κλέρ Ντέλη επίση για την υποχρέωση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν και την πυρηνική συμφωνία. Εκείνοι αποσύρθηκαν. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία είχε με τον προηγούμενο πρόεδρο της Αμερικής, τον Ομπάμα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το καταδικάσουμε τη στάση των ΗΠΑ δηλαδή. Ευχαριστώ. Χαμπίπ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πραγματικά ε, είμαι συνταραγμένος από την πρωινή συζήτηση. Ο μεγαλύτερος σύμμαχος ε, ε, το, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ιστορία και των κρατών της ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Όταν είπα πολύ σωστά επιβάλλουν κυρώσεις στο Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να υπονομεύσει αυτές τις κυρώσεις παγκοσμίω και μάλιστα δημιούργησε μια, ένα παράπλευρο τρόπο για να τις παρακάμψει και απέτυχε παρόλα αυτά. Τον Ιούνιο φέτος οι Ηνωμένε Πολιτείε ζήτησαν βοήθεια στα στενά του και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρισαν τα νότα τους στο αίτημα αυτό. Επίσης, ε, είχαμε την δέσμευση ενός πλοίου το, από το Ιράν και αυτό δεν θα είχε συμβεί αν δεν, είχε, αν ε, δεν είχαν υπονομεύσει οι Ευρωπαίοι τις αμερικανικές ε, δράσεις. Νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε το μεγαλύτερο σύμμαχο που είχαμε στην ιστορία. Ε, δεν βάζετε αρκετά χρήματα στο ΝΑΤΟ και παρόλα αυτά χρηματοδοτείτε ένα νέο αμυντικό ευρωπαϊκό σώμα. Είναι λάθος αυτό. Διορθώστε τις προτεραιότητές σας και συμπαραταχτείτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Ward, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ συνάντησα τον Ρίτσαρντ Ράτκλιφ, ε, τον σύζυγο της Ναζανίν Ράτκλιφ. Και μάλιστα για τρία χρόνια έκανε εκστρατεία για την αποφυλάξη της συζύγου του στο Ιράν. Έκανε και απεργία πείνα στις αρχές του έτους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη με την αδίκως φυλακισμένη σύζυγό του. Και μάλιστα η Ναζανίν βρίσκεται μόνη της σε μια χώρα που δεν αναγνωρίζει τη διπλή της ηθαγένεια και την ε, αναγκάζει σε απομόνωση στη φυλακή και μάλιστα έχει δεύτερη δίκη με πολύ πιθανή καταδίκη. Ε, είναι απάνθρωπος ο τρόπος κράτησής της και θα πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει. Η Ναζανίν είναι φυλακισμένη που, που μαζί με την Αράζα Ζαμίρη, Βρετανή Επίκο, ε, συνελήφθηκε, κρατείται από πέρυσι όταν επισκέφθηκε ε, την οικογένειά του. Καμίλα Μάντι επίσης, ε, σημαντικός ακτιβιστής ε, και ακαδημαϊκός από μη κυβερνητική οργάνωση που πρόσφατα συνελήφθη με άγνωστες καταγγελίες ε, στο Ιράν, άγνωστες κατηγορίες, δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ε, να τίθενται σε κίνδυνο η ζωή των ακτιβιστών. Επίσης ήταν παραπαλληλευτικέ και άτυχες ε, οι δηλώσεις του Μπόρι Τζόνσον όταν ήταν υπουργό Εξωτερικών. Νομίζω ότι αξίζουμε κάτι πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Με, με χαρά τώρα θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, η δέσμευσή μα για την υποστήριξη των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσων υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών είναι τμήμα τη πολιτική μα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώ σε πολλέ χώρε, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, οι γυναίκε εξακολουθούν να απειλούνται και να πέφτουν θύματα καταχρήσεων γιατί υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή γιατί απλούστατα είναι γυναίκε τις συκοφαντούν, τις μισούν, τις παρενοχλούν, τις εκφοβίζουν. Υφίστανται βία, σεξουαλικής φύσεως συχνά ή ποινέ φυλάκιση μόνο και μόνο γιατί περασπίζουν τα βασικά του δικαιώματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εκφράσω την βαθιά θλίψη μου προσωπικά για την Σαχάρα Κουνταγιάρη, η οποία νωρίτερα σε αυτό το μήνα αυτοπυρπολήθηκε όταν έμαθε ότι υπάρχει περίπτωση να φυλακιστεί μόνο και μόνο γιατί προσπάθησε να μπει σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο και πέθανε στο νοσοκομείο από τα τραύματά της. Είναι τραγικό μετά από την, τον όταν υφίστασε τέτοια περιφρόνηση, γιατί καμία γυναίκα δεν θα πρέπει να φυλακίζεται ή να φοβάται ότι θα φυλακιστεί μόνο και μόνο γιατί προσπάθησε να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Ε, έχουμε τη μέρα των γυναικών και όταν έρχεται αυτή τη στιγμή εμείς τιμούμε τις καθημερινές γυναίκες σε όλο τον κόσμο που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ιστορία μέσα στην χώρα τους και στις κοινότητές τους. Σε μια κοινή δήλωση που δημοσίευσε στις 8 Μαΐου η, γυναίκα, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος είπε ότι θέλουμε για όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια πρόσβαση στην υγεία, ε, στην εκπαίδευση, οικονομική άνεση για να διαμορφώσουν το δικό τους μέλλον. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να πολεμούμε για την πραγματική ισότητα για όλους εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλίσουμε ότι ό,τι έχουμε καταφέρει δεν ξεχαρβαλώνεται. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους ε, ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών και αυτό συμπεριλαμβάνει και το Ιράν. Στον πολιτικό διάλογο υψηλού επίπεδου που έχουμε τακτικά με το Ιράν, θέλουμε να προχωρήσουμε τη διμερή συνεργασία σε διάφορους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος και η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά θέτει το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτό το διάλογο. Έχουμε πολύ συχνά συζητήσεις ε, με τις αρχές για να ζητήσουμε οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και οι γυναικών, δεν θα πρέπει να είναι αντικείμενο παρενόχλησης, ε, βία κράτηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ε, το 2012 μάλλον, ε, μία γυναίκα η οποία πήρε και το βραβείο Ζαχάροφ, ε, καταδικάστηκε σε μακρές ποινές φυλάκισης και ήμασταν, εκφραστήκαμε κατά. Τα λέμε αυτά και στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το Νοέμβριο θα βγει το κείμενο για την κατάσταση στο Ιράν ε, και θα αναφέρουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Αγαπητοί Ευρωβουλευτέ, γνωρίζω ότι η εστίαση αυτή τη συζήτηση αφορά και την κατάσταση των υπηκόων με διπλή ηθαγένεια Ιράν και κάποια χώρα Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρακτική φυλάκιση ή κράτηση ατόμων όπως η Ναζανίν Ζαγκάρι Ράτκλιφ, ε, Βρετανο-Ιρανή, μόνο και μόνο λόγω της εθνικότητάς της, είναι εναντίον του Παγκόσμιου Συμφώνου για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα που επικύρωσε το Ιράν και δεσμεύεται λοιπόν να τηρήσει. Η συνεχής πρακτική κράτησης αυτών των ατόμων με διπλή ηθαγένεια παραβιάζει τη δέσμευση ότι κανένας δεν θα υφίσταται αυθαίρετες συλλήψεις ή κρατήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να ζητούμε την απελευθέρωση όλων των υπηκών με διπλή θαγένεια Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιράν και των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμε από το Ιράν επίσης να εξασφαλίσει την απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται αυθαίρετα και ότι οι φυλακισμένοι δεν θα την χάνουν κακομεταχείρισης. Οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο που τον επιλέγουν οι ίδιοι και επαρκεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ξανατονίζω ότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και μας δίνει θάρρος η σημασία που δίνουν οι Ευρωβουλευτές στο θέμα αυτό. Δεν θα αφιστούμε κόπον, ούτω ώστε να υποστηρίξουμε τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επιτροπέ. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος για να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή από τις εξή πολιτικές ομάδες. ECR, Πράσινη, ε, Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία, S&D, Renew, GU, NGL και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, κλείνει η συζήτηση, η ψηφοφορία θα γίνει αργότερα. Διακοπή μέχρι τις ψηφοφορίες στις 12 ακριβώς. Επάναλαμβάνετε Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ καθίστε. Από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο πρόεδρο ε, έλαβε την εξή απόφαση για αλλαγή ορισμού σε μία αντιπροσωπεία. Ο κύριο Γιώζα Ολέκα. Ε, θα ε, συμμετάσχει στην κοινοβουλευτική διάσκεψη Euronest στη θέση του κυρίου Σβέν Μίξερ. Η απόφαση αυτή ε, τίθεται αμέσως σε ισχύ την ίδια μέρα της ανακοίνωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχαμε μια μικρή καθυστέρηση γιατί διήρκησε λίγο περισσότερο η διάσκεψη των Προέδρων και μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε είναι οι ακροάσει των Επιτρόπων σημαντικές για όλους μας και άκουσα ότι η διάσκεψη των Προέδρων τώρα τελείωσε και δεν είναι πολύ μακριά για να έρθουν με τα πόδια. Θα ήθελα επευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους σας, ιδιαίτερα στους νέους βουλευτές και να πω ότι πάντα στις τελευταίες ψηφοφορίες έχουμε συναδέλφους που βιάζονται την τελευταία μέρα και πολλές φορές οι συνάδελφοι όταν ψηφίζουν ξεχνάνε την κάρτα τους στο μηχάνημα. Αχ, πηγαίνετε να φέρετε τη δική μου κάρτα, σας παρακαλώ γιατί είναι στο έδρανό μου. Λοιπόν, ε, μην, βγάζετε τις κάρτες σας αμέσως πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία ηλεκτρονική, γιατί βιάζεστε να φύγετε, γιατί έτσι αποσύρετε και την ψήφο σας και όταν είναι ομαστική ψηφοφορία δεν θα φαίνεται στα πρακτικά. Ε, πράγμα που έχει σημασία και για άλλες διαδικασίες. Λοιπόν, παρακαλώ, ακόμα και αν πρέπει να φύγετε, να μην βγάζετε την κάρτα από τη σχισμή μέχρι να ανακοινωθεί ότι ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ε, ήρθε ο πρώτος πρόεδρος πολιτικής ομάδας ήδη, αλλά μάλλον οι πράσινοι έρχονται τρέχοντας. Βλέπω να καταφθάνουν και άλλοι για να αρχίσουμε τις ψηφοφορίες. Η πρώτη ψηφοφορία δεν είναι ονομαστική και αρχίζουμε με την κατάσταση στην Τουρκία, ιδιαίτερα με την καθαίρεση των ερετών δημάρχων. Ε, πρώτα το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι το ψήφισμα του ECR. Ερχόμαστε στο κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Είναι η τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Αρχίζει τώρα παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3, ονομαστική κλίση, αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Abgelehnt. Απορρίπτεται. Η, η τροπολογία 1D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το σύνολο του ψηφίσματος, όπως δεν τροποποιήθηκε, ψήφι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτουν τα υπόλοιπα ψηφίσματα. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα για τη Μιανμάρ, Βιρμανία, ιδιαίτερα την κατάσταση των Ροχίνγκια. Έξι πολιτικές ομάδες έχουν καταθέσει ε, ψήφισμα τροπολογία 1, υπέρ κατά, μετά την αιτιολογική σκέψη H, αποχές απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές. Μάλλον έχει εγκριθεί, αλλά βλέπω πολλές αποχές. Παρακαλώ να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεν βλέπω. Όχι, όχι, έχει πολλέ αποχέ. Ε, λοιπόν, το επόμενο ψήφισμα. Η Ιράν, ιδίω η κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν τη διπλή ηθαγένεια. Ευρωπαϊκή Ένωση Ιράν. Ένα ψήφισμα από πέντε πολιτικέ ομάδε. Η τροπολογία 2 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, η τροπολογία 1 και πάλι ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 ψήφι κατά απόχες απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στο ψήφισμα σχετικά με τη δυνατότητα κατοχήρωση φυτών και κατοσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Είναι από έξι πολιτικές ομάδες. Συνεχίζουμε το ψήφισμα για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Παράγραφος 3, το αρχικό κείμενο ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Εδώ ε, έχει ζητηθεί προφορική τροπολογία που θα την παρουσιάσει ο συνάδελφος Φεστ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ένα ψήφισμα ε, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, για την μνήμη. Οκτώ σελίδες μιλάει για τον ολοκληρωτισμό, για διάφορα πράγματα, αλλά πουθενά δεν αναφέρει τους Εβραίους. Λες και δεν θανατώθηκαν αυτοί, αλλά οι Ρωμά, μειονότητες, ο πρόεδρος δεν θα κάνετε αιτιολόγηση. Μήπως να μας παρουσιάζατε την προφορική σας τροπολογία. Αυτή τη στιγμή δεν χωράνε περισσότερα. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Φέστη. Δεν φταίει ο συνάδελφος, εγώ του έκλεισα το μικρόφωνο. Ε, ανάψτε το και πάλι. Έλεγα λοιπόν, ε, στο 4 έχουμε μια ε, προφορική τροπολογία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκφράζει το βαθύ σεβασμό και τώρα έρχεται η τροπολογία προς τα εκατομμύρια ε, των Εβραίων θυμάτων του ολοκαυτώματος που οδήγησε στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ και όλα τα υπόλοιπα θύματα κτλ. Και να παρακαλέσω όλους τους αντισημίτες εδώ ε, πράσινους, σοσιαλδημοκράτες και γκουε. Για σηκωθείτε υπέρ της δικής μας τροπολογίας για να δούμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Συνάδελφε, ήδη στην αρχή σας έκοψα το λόγο. Αυτό τα τελευταία ήταν περίτα. Στο μέλλον, αν το ξανακάνετε, θα σας ανακαλώ στην τάξη. Ο συνάδελφος Μελχιόρ στο 732 η κυρία Μελχιόρ. Διαδικαστικό έχετε. Διαδικαστικό. Οι διερμηνείς δεν προσλαβαίνουν να μεταφράσουν τον ομιλητή πριν το πέρας των ψηφοφοριών. Οπότε οι Γερμανοί, οι γερμανόφωνοι καταλαβαίνουν τι ψηφίζουμε. Γιατί άκουσαν το πρωτότυπο, αλλά οι υπόλοιποι από τη στιγμή που δεν προλαβαίνουν οι διερμηνήσεις δεν καταλαβαίνουμε το περιεχόμενο. Θα πρέπει οι ομιλητή να μιλούν λίγο πιο αργά. Also, Frau Kollegin, lassen Sie uns... Αγαπητέ συνάδελφοι, ένα-ένα τα θέματα σας παρακαλώ. Πρώτα έχουμε την τροπολογία αυτή την προφορική του κυρίου Φέστ και ονομαστική ψηφοφορία που θα γίνει. Αλλά ερωτώ, διαφωνεί κανείς? με την προφορική αυτή τροπολογία. Das Από ό,τι φαίνεται όχι. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Meine Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε ακόμα νεαρό κοινοβούλιο. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να κάνουμε προφορικές τροπολογίες. Το επιτρέπει ο κανονισμός. Στη συνέχεια δεν γίνεται συζήτηση, ούτε ζητεί κανεί το λόγο, απλώ ρωτάει ο πρόεδρο. Αν διαφωνεί κανεί, να κατατεθεί η προφορική τροπολογία. Και αν εγερθούν 40 συνάδελφοι, τότε δεν ψηφίζεται η προφορική τροπολογία. Αν δεν εγερθούν 40 συνάδελφοι, ψηφίζεται η τροπολογία χωρίς συζήτηση περαιτέρω όμως. Συνάδελφε, για να είμαστε δίκαιοι, κύριε Χέρψ. Äh, Κύριε Φεστ και όχι Χέρμπστ. Κύριε Φεστ. Ναι, βάλτε ακουστικά αν δεν με ακούτε, παρόλο που μιλάμε την ίδια γλώσσα. Κύριε Φεστ. Συμφωνείτε να σας ρωτήσω δεύτερη φορά ποιος έχει αντιρρήσεις κατά της προφορικής τροπολογίας. Οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ακόμα όλες τις διαδικασίες. Ο συνάδελφος Φέστ θεωρεί ότι δεν είναι δίκαιο και σωστό να ρωτήσω δύο φορές, οπότε ας ψηφίσουμε την τροπολογία αυτή. Ονομαστικά. Ονομαστική ψηφοφορία. Ε, την επέτρεψα και θα την κάνουμε. Έκανε μια προφορική τροπολογία ο συνάδελφος και ταυτόχρονα ζήτησε και ονομαστική ψηφοφορία. Και το επιτρέπω. Τώρα έχει έρθει και ένα διαδικαστικό. Ποιος το ζήτησε, ο κύριος Κοβάτσεφ. Ε, Με εξέπληξε αυτή η κατάσταση. Συνήθως η ονομαστική ψηφοφορία ε, και το σχετικό αίτημα θα πρέπει να γίνεται αρκετές μέρες πριν είναι δυνατόν να ζητήσει κανεί ε, ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία τη στιγμή που υποβάλλει το αίτημα για προφορική τροπολογία και μάλιστα να το δεχτείτε. Κοιτάξτε, συνάδελφε Κοβάτσεφ, τα τελευταία τρία χρόνια έχω μελετήσει σχολαστικά τον κανονισμό και ομολογώ ότι το ξέρω 100% απ' έξω. Αλλά δεν γίνεται να ζητήσει κάποιος τέσσερις μέρες πριν ε, ονομαστική ψηφοφορία όταν κάνει προφορική τροπολογία τη στιγμή της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι ήταν μια αυθόρμητη, σωστή απόφασή μου να πω αν δεν διαφωνεί κανείς με την προφορική τροπολογία να γίνει ονομαστική ψηφοφορία και να το τηρήσουμε ενιαία. Έτσι το αποφάσισα εγώ και θα γίνει κιόλας. Αρχίζει τώρα η ονομαστική ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η τροπολογία. Gibt es noch Wortmeldungen? Θέλει κανείς το λόγο ε, για θέματα που δεν έχουν ε, διεκπεριωθεί από την ψηφοφορία. Όχι, η αρχική παράγραφος 6 ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 12 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο, ονομαστικά παρακαλώ, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην παράγραφο 20. Έχουμε την τροπολογία υπαριθμένα και εδώ προφορική τροπολογία του κυρίου Μπιουτικόφερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για την τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών έχουμε μια προφορική τροπολογία εμείς να σας τη διαβάσω στα αγγλικά. Ε, η τροπολογία των σοσιαλιστών και δημοκρατών προσθέτει τα εξής και παραθέτω. Και να απαγορευτούν ε, αποτελεσματικά νεοφασιστικές και νεοναζιστικές ομάδες και οποιαδήποτε άλλα ιδρύματα ή ενώσεις που υμνούν ε, ή δοξάζουν τον ναζισμό και τον φασισμό. Και εδώ ζητώ να προσθεθεί προφορικά ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ολοκληρωτισμού. Ευχαριστώ πολύ. Διαφωνεί κανείς κατά της προφορικής αυτής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν Μέχρι τώρα μετράω 24 συναδέλφους, αν μέτρησα σωστά. 40 απαιτούνται, οπότε θα ψηφίσουμε την αρχική ε, τροπολογία επαριθμών 1 με την τροποποίηση που έγινε από την προφορική τροπολογία και μάλιστα ονομαστικά. Αρχίζει τώρα λοιπόν η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρασε. Εγκρίνεται. Και ερχόμαστε στην ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Κυρίε και κύριοι, ερχόμαστε τώρα στο επόμενο ψήφισμα για την κατάσταση τη εφαρμογή νομοθεσία για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε για το ξέπλεμα. τέσσερι πολιτικέ ομάδε έχουν καταθέσει ψήφισμα. Ονομαστικά ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 2 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 και πάλι ονομαστικά αρχίζει η ψηφοφορία. Αν ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 4 ονομαστικά αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος, θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η κυρία Μελχιόρ για το ρυθμό και την ταχύτητα. Προσπαθούμε ε, όσο γίνεται να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ε, με γοργούς ρυθμούς. Πάντα στην αρχή της θητείας ε, σημειώνουμε ότι οι συνάδελφοι διαμαρτύρονται ότι τα λέμε πολύ γρήγορα και στο τέλος της θητείας ότι τα λέμε πολύ αργά. Σας διαβεβαιώ ότι εγώ έχω αυτό το ρυθμό και μάλιστα τον έχω μειώσει λίγο τον κανονικό μου ρυθμό. Και είμαι βέβαιος ότι και με όλους τους άλλους αντιπροέδρους και με μένα τελικά κάπως θα συντονιστούμε και θα τα βρούμε. Το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστικά αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Σε όσους φεύγετε καλή επάνωδο, καλό ταξίδι. Και όπως πάντα θέλω να παρακαλέσω θερμότατα τους συναδέλφους να φύγουν γρήγορα από την αίθουσα όσοι θέλουν να αποχωρήσουν έτσι ώστε να ακούσουμε εκείνους που θέλουν να κάνουν επεξηγήση ψήφου και ενδιαφέρονται να ακούσουν τις επεξηγήσεις αυτές απρόσκοπτα. Α,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 der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, liebe Λοιπόν, κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα αναφέρω ονόματα τώρα, Κασπάρη, για όσου μιλούν στου διαδρόμου. και Σάγερ. Ins Protokolleingang. Και σα γράφουμε και στα πρακτικά. Der Herr Kollege Hennen beschäftigt auch drei Kollegen. Και ο κύριο Χάναν Απασχολεί τρεις συναδελφούς που θέλουν να φύγουν. Die Frau Κυρία Άουκεν, κυρία Νιτφέλτ, ο κύριος Μπιτικό, φέρω όλα τα πηγαδάκια. Herr Kollege Gahler, genau. Α, και εσείς κύριε Γκάλερ, ναι, ναι, ακριβώς. Herr Kollege Liese, Herr Kollege Linz, Herr Kollege Kovacev. So, wir haben insgesamt... Λοιπόν, έχουμε συνολικά 20 επεξηγήσεις ψήφου. Αρχίζουμε με το ψήφισμα που αφορά τη δυνατότητα κατοχήρωση φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα έβρεση τεχνίας. Κυρία Σόεντροβα, μισό λεπτό κυρία Σόεντροβα. Εδώ είμαι. Ναι, αλλά περιμένετε λίγο. Ζητώ συγγνώμη. Könnten Παρακαλώ εκεί στη δεξιά πτέρυγα, λίγο ησυχία. Κυρία Σόιντροβα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε στη δυνατότητα κατοχύρωσης ε, των φυτών ε, και βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρυστεχνίας. Νομίζω ότι ήταν σαφέ το μήνυμα που στείλαμε στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφευθεί οποιαδήποτε νομική επιπλοκή. θα πρέπει να έχουμε νομική σαφήνεια, ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα κατοχήρωσης με δίπλωμα ευρυστεχνίας ε, φυτών και βιολογικών διεργασιών. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφές ε, στο Συμβούλιο ε, Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρυστεχνίας. Και απευθύνουμε και έκκληση προς τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να συνδράμουν ώστε να διαλευκανθεί η νομική κατάσταση, γιατί υπάρχει έλλειψη ασφαλής δικαίου. Ευχαριστώ κυρία Σόδροβα. Παρακαλώ, εσείς εκεί, οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές, όλη η ομάδα, σας παρακαλώ αν θέλετε να αποχωρήσετε, να το πράξετε ταχαίως, συνάδελφοι. Please, colleagues, it would be very polite. Συνάδελφοι, νομίζω ότι ήταν πολύ ευγενικό να εγκαταλείψετε αμέσω την αίθουσα τη Ολομέλεια. Ε, Αλλιώ ε, καθίστε παρακαλώ. So, thank you. Ευχαριστώ κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί υπερψήφισα. Η δυνατότητα κατοχήρωσης φυτών και κατ' ουσία βιολογικών διεργασιών με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να γίνεται υπό όρους, να υπάρχει δυνατότητα κατοχήρωσης ή κατοχήρωση πνευματικών και συγγενών δικαιωμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το γενικό συμφέρον σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο πολλαπλασιαστικό φοιτικό υλικό. Για όλους αυτούς τους λόγους υπερψήφισα το ψήφισμα, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και να απευθύνομαι προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευχαριστώ κυρία Ρίτσι. Ευχαριστώ. Το θέμα της δυνατότητας κατοχήρωσης ζωντανών οργανισμών ε, με συγκλώνησε, με σόκαρε. Φαίνεται ότι είμαι πολύ αφελής. Είναι δυνατόν ε, ε σπόρους ή πολλαπλασιαστικό υλικό που κανονικά πρέπει να ανήκουν στη δημόσια γνώση να το μετατρέπουμε σε γνώση μόνο πολυεθνικών που θα κατοχυρώνεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνία, τέτοια γνώση θα πρέπει να είναι προσιτή σε μικροκαλλιεργητέ και βελτιωτέ φυτών. Η δυνατότητα καταχύρωση φυτών και βιολογικών διεργασιών. Εκτός ότι κάνουν τις πολυεθνικές να, μονομελούν τη γνώση, από, να μονοπολούν τη γνώση απομονώνοντα του καλλιεργητέ, αποβαίνει και ει βάρο των δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, γιατί πλήττει τα τοπικά οικοσυστήματα και τη δυνατότητα και κάποιων κρατών να έχουν την κυριαρχία της επιστηστικής ασφάλειας. Ουσιαστικά μεγάλες πολυεθνικές ε, κλέβουν τη γνώση των εθνικών φυτών που για πολλές γενιές την είχαν οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Γιατί ο μόνο τρόπο για να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη γνώση τελικά οι καλλιεργητέ είναι να την αγωνάζουν από τι πολυεθνικέ, αν το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ, συνάδελφο Ολέκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ποικιλία των φυτών είναι πηγή για την ανάπτυξη νέων φυτικών ειδών. Αυτή η ποικιλία, η φυτική ποικιλία, δεν αρκεί όμως για να αναπτυχθούν νέα είδη και να προστατευτεί η βιοποικιλότητα. Πρέπει να υπάρξει και καινοτομία παράλληλα. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και σε αυτή την κατέθεση και αυτό είναι σημαντικό για την παραγωγή τροφίμων. Η κατοχήρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνία είναι σημαντική μερικέ φορέ. Ο κάτοχος του διπλώματο δεν θα δώσει πάντα την, τους πόρους του παραδείγματος χάρη δωρεάν. Θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για να ξέρουμε πότε οι σπόροι μπορεί να δοθούν ας πούμε, σε άλλον. Δεν θα πρέπει οι καλλιεργητές να βασίζονται στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να κάνουν τη δουλειά τους. Και πιστεύω ότι δεν μπορούμε να εκδίδουμε ε, διπλώματα ευρεσιτεχνίας για γενετικό υλικό. Ευχαριστώ, κύριο Χάναν. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Η πρόοδος στην, στην δημιουργία φυτών και στην καλλιέργεια φυτών γίνονται όλο και καλύτερα έχουμε μεγαλύτερη απόδοση από μικρά αγροτεμάχια. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι μόνο ότι μπορούμε να θρέψουμε τον κόσμο ε, με έναν τρόπο που μια γενιά πριν θα ήταν αδιανόητο, όχι μόνο ε, όλες τις προβλέψει ικτρές ε, ε, προβλέψεις και τους κασανδρισμούς ότι θα πεινάσουμε τις έχει διαψεύσει, αλλά μπορούμε έτσι να επιτρέψουμε την ανανέωση ε, προηγουμένως επαπειλούμενων ε, ειδών ε, και την ανανέωση των δασών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι προπομπός αυτής της τεχνολογίας. Συχνά ένας συνδυασμός όμως και εκτιμένων συμφερόντων και κακών πολιτικών μας αποκόπτουν από την πρόοδο στο, στη γενετική επιστήμη. Ελπίζω εμείς οι Βρετανοί να είμαστε προπομπή ε, σε αυτό το πεδίο, αλλά ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ κύριε Χάναν. Προχωρούμε στα υπόλοιπα ψηφίσματα. Και επόμενο είναι η σημασία της Ευρωπαϊκής Μνήμης για το μέλλον της Ευρώπης. Η κυρία Μπίλντα έχει πρώτη το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η το ψήφισμα, το οποίο δεν είναι αμερόληπτο, δεν νομίζω ότι τιμάει τα θύματα του ολοκληρωτισμού. Καταρχάς, ε, η μνήμη του τελευταίου παγκόσμιου πολέμου ε, δεν θα πρέπει να γίνεται όμοιρος πολιτικών συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν θα πρέπει να πέφτει σε λαϊκισμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τη στιγμή που γίνονται διάφορες εκλογές και ο κόσμος πηγαίνει προς πιο ακραίες τάσεις, θα πρέπει εμείς να κατοχυρώσουμε την ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο... Όταν υπάρχει άρνηση της ιστορίας ε, μέσω αυτών κειμένων, δεν νομίζω ότι θα τιμήσει τους 20, τα 20 εκατομμύρια ε, Ρώσων που θυσιάστηκαν για να ζήσει η Ευρώπη. Ε, ξαναγράφεται ιστορία με αυτό το ψήφισμα που υποτίθεται ότι καταγγέλει τα δικτατορικά καθεστώτα. Διερωτώ με, τι φύση ε, αποκτά αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γινόμαστε όλο και πιο, α, αλλάζουμε πρόσωπο. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αξιότιμοι, Αξιότιμοι συνάδελφοι. Εγώ υπερψήφισα το ψήφισμα γιατί πιστεύω στην ιστορική μνήμη. Όπως και άλλα αντιδημοκρατικά καθεστώτα, ε, ας μην ξεχνούμε και την πολσεβικική καταπίεση. Ζήσαμε κάτω από την βότα των πολσεβίκων στην Ευρώπη για μία πεντηκονταετία. Θα ήθελα να σας δώσω ως παράδειγμα την απόπειρα που έγινε να διχαστεί το βουλγαρικό ε, έθνος και να δημιουργηθεί η μακεδονική οντότητα στο βουλγαρι... στη βουλγαρική επικράτεια. Τέτοιου είδους ε, ε, βαρβαρότητες θα πρέπει να καταδικαστούν και η αυταρχικότητα του σφυροδρέπανου. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, ο συνάδελφος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος. Είμαι από τους λίγους ευρωβουλευτές που γεννήθηκαν εξόριστοι. Εκπροσωπούμε τον ευρωπαϊκό λαό και έχουμε καθήκον να διεκδικούμε καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη. Τίποτα καινούργιο δεν υπάρχει. Πριν από 80 χρόνια τις ίδιες ελπίδες είχαν και οι παππούδες μας. Αλλά οι τύρανοι, οι δεσπότες υπονόμευσαν αυτή την προσδοκία υπογράφοντας μυστικά πρωτόκολλα και συμφωνίες ε, που προκάλεσαν μεγάλες ε, μετακινήσεις στο ολοκαύτωμα και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μαζί με άλλες δεκάδες χιλιάδες Λιθουανούς, οι γονεί μου ε, σε τρένα μεταφορά ζώων εξορίστηκαν στη Σιβηρία. Εγώ εκεί γεννήθηκα. Και δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο δώσαμε τη μάχη για την ελευθερία μας. Όπως βλέπουμε στην αίθουσα αυτή, ένα τμήμα των Ευρωβουλευτών φαίνεται ότι αγνοούν την ιστορία, αγνοούν την κατάσταση πέρα από το σιδηρού παραπέτασμα ε, το παραπέτασμα. Θα πρέπει λοιπόν, ε, αν θέλουμε μια δικαιότερη Ευρώπη για τα παιδιά και τα εγγόνια μας, να αποτρέψουμε την επανάληψη της ιστορίας στο μέλλον. Ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή. Η κυρία Φόξ έχει το λόγο, παρακαλώ. resolution. Εγώ καταψήφισα όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει η ιστορική μνήμη, αλλά με πάρα ενδιαφέρουν τα ιστορικά γεγονότα και η μνήμη. Γι' αυτό δεν θέλω να μετατρέψουμε ε, ένα, την ιστορία σε ένα ρεβιζιονιστικό ποδόσφαιρο. Ε, γιατί μερικές φορές ε, αντιμετωπίζουμε ε, με περιφρόνηση και ισοπεδώνουμε την ιστορία. Γιατί δεν μιλούμε για τον γιατί φαίνεται ότι εξομοιώνουμε ε, το φασισμό και το ολοκαύτωμα και τα δεινά των ε, ε, Εβραίων με κάποιες προσπάθειες φεντεραλισμού και επεκτατισμού. Έχουμε το διαφωτισμό, την αναγέννηση, τις τέχνες δεν θα, θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Έχουμε την αυτοδιάθεση, τα κράτη-έθνη, την εθνική κυριαρχία, τη δημοκρατία. Αυτέ είναι οι αρχέ που φαίνεται να ξεχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τι αψηφά. Εγώ όμω τι θυμάμαι και γι' αυτό καταψήφισα το σχετικό ψήφισμα που δεν είναι παραπολιτική προπαγάνδα. Ευχαριστώ κύριε Φόξ. Ο συνάδελφο Πάλμερ. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Είμαι αυτή μία από τις πιο σημαντικές, τα πιο σημαντικά κείμενα που εγκρίθηκαν σήμερα. Εξασφαλίζουμε στους νέους και στις μελλοντικές γενιές τη γνώση για το τι συνέβη στις πιο σκοτεινές σελίδες της ε, ιστορίας της, Ευρωπαϊκής, της Ευρώπης. Ε, είναι πολύ σημαντικό, καταρχάς, ε, ε, το Μουσείο Ολοκαυτώματος ε, στα Μίτλαντ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι μαθητές, οι νέοι, καταλαβαίνουν τι, συνέβησε, τι συνέβη τότε. Και καταλαβαίνουν και το ρόλο τους και μπορούν να σταματήσουν το μίσος και τις ρητορίες μίσους. Θέλω να τιμήσουμε τους, τα θύματα του Ολοκαυτώματος ε, και θα πρέπει όλοι μας σήμερα και οι νέοι να καταλάβουμε τι συνέβη τότε και να έχουμε τα εργαλεία ούτω ώστε όταν λέμε ποτέ πια να σημαίνει πραγματικά αυτό που λέμε ποτέ πια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Βίντσε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη πρέπει να θυμάται ούτως ώστε οι φρικαλαιότητε που συνέβησαν στον 20ο αιώνα να μην ξανασυμβούν ούτε ο φασισμός ούτε ο κομμουνισμός. Οι χώρες της Κεντρική και ανατολικής Ευρώπης ε, αντιμετώπισαν ε, και φασισμό και κομμουνισμό τα περασμένα χρόνια, τις περασμένες δεκαετίες. Ε, η γενιά μου επηρεάστηκε ε, εν μέρη από την δικτατορία στη Ρουμανία, αλλά πολύ περισσότερο γενιά του πατέρα μου και του παππού μου. Οι ιστορικές εκκλησίες καταστράφηκαν και δεν έχουν αποκατασταθεί, παρότι υπάρχει νόμος που απαιτεί από το κράτος να τις αποκαταστήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε στις κρατικές αρχές ότι πρέπει να εφαρμόσουν το δίκαιο. Στην κεντρική Ευρώπη υπάρχει μια καθυστέρηση 50 ετών σε ό,τι αφορά την οτροπία τα ταμεία συνοχής εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το θέμα. Ε, πρέπει να προσπαθούν να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα. Η ιδέα ποτέ πια είναι κάτι που πρέπει να περάσουμε ως λαμπάδα σε επόμενες γενιές. Ευχαριστώ, συνάδελφος Χουκ. Χαίρομαι που μπόρεσα να υποστηρίξω αυτό το ψήφισμα για να θυμόμαστε τα θύματα του ολοκληρωτισμού. Για μας είναι και προσωπική ιστορία. Οι παππούδες της γυναίκας μου ήταν επιζώντες του Auschwitz, του Auschwitz και με αγγίζει ως το μεδούλι που τα πράγματα θα μπορούσαν να, να είναι τελείως διαφορετικά και στο τσακ γεννήθηκε η γυναίκα μου και τα παιδιά μου λοιπόν. Ε, οι παππούδες μου α, έφυγαν με τρένα την ώρα που πέφτανε ε, βόμβες από τον ουρανό. Η, μας ενώνει η ιστορία μας τους Ευρωπαίους και η μνήμη και είμαστε αποφασισμένοι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά παρά μια επιφύλαξη που έχω, υπερψήφισα το ψήφισμα. Ε, το πρόβλημα είναι ότι το ψήφισμα μιλάει για τη φρικαλαιότητα Ευρωπαίων αντίον άλλων Ευρωπαίων. Όμως ε, έχουν σημειωθεί φρικαλαιότητες και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε Ευρωπαίους σήμερα που οι πρόγονοί τους έρχονται από την Αμερική, την Αφρική και την Ασία. Όλες οι φρικαλαιότητες πρέπει να τις τιμόμαστε και να τιμούμε όλους τους προγόνους από όπου και αν προέρχονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουκ. Δεν βλέπω το συνάδελφο Τέρτς, οπότε θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χάναν. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Πριν 80 χρόνια, μισό εκατομμύριο ε, ε, στρατιώτες του το, κόκκινου στρατού ε, μπήκαν στην Πολωνία ε, μαζί με αεροπλάνα κτλ. σε μια μαζική επίθεση. Δημιουργήθηκε η ιστορία ότι βοήθησαν τους Σλάβους αδελφούς εναντίον των Ναζί, αλλά ξεκαθαρίστηκε η πρόθεσή τους. Στην πραγματικότητα, Σοβιετικοί και Ναζί, οι στρατηγοί ε, έφαγαν μαζί και κάλεσαν τους ε, Ναζί να τους επισκεφτούν στη Μόσχα μετά. Ε, υπάρχει επιλεκτική αμνησία εδώ που τμήμα της σημερινής μοντέρνας αριστεράς για την συμφωνία αυτή είναι εντυπωσιακό και δείχνει την τρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας λένε ότι ο κόκκινος στρατός μας απελευθέρωσε, ότι απλώς η Δύση ε, λιγάκι βοήθησε ας πούμε. Ε, αλλά ξέχασαν ότι περίπου για το 1 τρίτο της, του πολέμου ήταν η Σοβιετικοί στο πλευρό των Ναζί. Ευχαριστώ κύριε Χάναν. Η κυρία Σδενόκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα. Παρόλο που ήμουν υπέρ κάποιων παραγράφων του ψηφίσματο. ήμουν κατά της συνολική προσέγγιση που εξομοιώνει το σναζί με το κομμουνιστικό καθεστώς. Ε, το κακό είναι μόνο ένα και ο απόλυτο σατανά είναι η ναζιστική ιδεολογία. Είμαι κατά της ποινικοποίηση τη ε, προσέγγιση της ιστορίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που κάτι που κάνει το ψήφισμα. Τι έγινε με το Μόναχο, το ξεχάσαμε. Τι γίνεται με τις διμερείς συμφωνίες που συνάφθηκαν πριν, πολύ πριν τις 28 Αυγούστου του 1939. Η δική μου οικογένεια θυσιάστηκε, υπέφερε από τους Ναζί και ε, υπέφερε από τη μετακίνηση, από τον εξορισμό, αλλά ο σατανάς είναι ένας και ο σατανάς είναι η ναζιστική ιδεολογία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σντανόκα. Τελευταία η κυρία Γουόρντ, παρακαλώ. Ε, thank you. Ευχαριστώ. Ω μέλο τη Επιτροπή Παιδεία και Πολιτισμού την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και τώρα ω αντιπρόεδρο τη ίδια Επιτροπής ανέκαθεν προσπαθώ να μιλήσω για την ανάγκη ιστορική μνήμη. Δύσκολη ιστορία, είτε μέσω του το του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη ή το, της Δημιουργικής Ευρώπης. Είμαι εδώ γιατί ο, Κένι Τσάπλιν, ο ανυψιός της μου, βρίσκεται ε, στη Νότια Γαλλία ε, Το 1918 δολοφονήθηκε ε, στον αγώνα του κατά το φασισμό. Η Ευρωπαϊκή, κατά φασισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φιλιρινικό σχέδιο, γιατί η, Ευρωπαϊκή, η Ευρώπη δεν, μπορεί, δεν έχει την πολυτέλεια άλλου πολέμου. Είναι τεράστιο το ανθρώπινο κόστος και είχαμε μαζικές εκτοπίσεις και δεινά σε όλη την Ευρώπη. Εμείς κάνουμε μια κοινή προσπάθεια με συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών να δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό όραμα. Και αυτό το σημείο καμπή ε, του προηγούμενου αιώνα θα πρέπει να το ε, διηγηθούμε και να ε, γύρουμε την ευαισθητοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Θέλουμε ανοχή, αμοιβαία κατανόηση και επανασυμφιλίωση. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε και με το ψήφισμα αυτό και ερχόμαστε στις επεξηγήσεις ψήφου σε σχέση με την κατάσταση της εφαρμογής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η κυρία Σόιτροβα. Υποστήριξα αυτή την πρόταση ψηφίσματος για να εφαρμοστεί η νομοθεσία, για να καταπολεμηθεί η νομιμοποίηση εσόδων. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό Έχουμε τα έγγραφα του Παναμά. Ξέρουμε τι αγώνας διεξάγεται για την καταπολέμηση ε, τέτοιων εσόδων. Έχουμε 10 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες που δεν εφάρμοσαν την οδηγία για την καταπολέμηση των εσόδων αυτών. Και χαίρομαι που η χώρα μου, η τσεχική δημοκρατία, δεν ανήκει σε αυτές τις 10 χώρες. Πρέπει να τονίσουμε ότι αυτή η νομοθεσία είναι σημαντικό και πρέπει να εφαρμοστεί θα πρέπει όλα τα τραπεζικά συστήματα να συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες για αυτό. Δυστυχώς, το ξέπλυμα χρήματος δεν έχει σύνορα. Ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμιο επίπεδο για να την καταπολεμήσουμε. Ευχαριστώ κυρία Ομπχή παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό είναι σημαντικό το 1% του ΑΕΠ στην Ευρώπη ενέχεται σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Είναι αντίστοιχο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ε, οι φοροδιαφεύγοντες εκμεταλλεύονται αυτά τα τραπεζικά παραδειράκια. Θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε ότι είμαστε δύναμοι ως Ευρωπαϊκή Ένωση να επεμβαίνουμε. Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή έδειξε πόσο ανίκανη είναι και αδύναμη, δεν έχει επιβάλει καμία κύρωση. Έχω υπογράψει το ψήφισμα αυτό, το διακομματικό και ελπίζω να είναι μια σημαντική φάση ε, στον αγώνα των, ε, της ενίσχυσης των μέσων κατά του ξεπλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αλλά δεν θα γίνει αυτό αν δεν έχουμε ένα κατάλογο εξαντλητικό των φορολογικών παραδείσων, γιατί είναι διαβόητη κάποια φορολογική παράδοση που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν δεν το κάνουμε αυτό, είμαστε καταδικασμένοι να αποτύχουμε. Ευχαριστώ κυρία Ομπρή. Δεν βλέπω τον συνάδελφο Μορέλ, ούτε τον συνάδελφο Πόλτσακ ε, στην αίθουσα. Ε, τελευταίος, ο κύριος Τζαμπάσκι, παρακαλώ. Εγώ ψήφισα αποχή. Φυσικά και είμαι κατά του ξεπλήματο χρήματο, κατά τη νομοποίηση παράνομων εσόδων, αλλά κάποια στοιχεία του ψηφίσματο ε, νομίζω ότι σεβετερίζονται τι εθνικέ αρμοδιότητε. Μιλούμε για τον ΑΒ οργανισμό που μπορεί να καταπολεμήσει το πρόγραμμα, αλλά δεν νομίζω ότι η γραφειοκρατία ή η σύσταση ενό νέου οργανισμού θα είναι η λύση. Όχι, είμαι κατηγορηματικός. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θα πρέπει να τηρούμε την νομοθεσία και να μην τις χρησιμοποιούμε ως ε, μέσο για να, για να υλοποιήσουμε τους πολιτικούς μας στόχους και να ε, στυλιτεύσουμε κάποιες χώρες, στην περίπτωση αυτή την Ουγγαρία και την Πολωνία. Ευχαριστώ κύριε Τζαμπάσκη. Τελείωσαν οι επεξηγήσεις ψήφου και για αυτό το ψήφισμα, για το ξέπλυμα και εξαλίσαμε και την ημερήσια διάταξη. Σας εύχομαι ένα ευλογημένο γεύμα και διακόπτω τη συνεδρίαση μέχρι τις 3.